Καλημέρα συνάδελφοι, σας παρακαλώ καθίστε. Φτάνει ο Επίτροπος, έφτασε μάλλον. Οπομένως μπορούν να αρχίσουν οι εργασίες μας σχεδόν στην ώρα μας. Με μεγάλη χαρά υποδεχόμαστε όλοι μας τον Επίτροπο Όλη Ρεν. ήταν πολύ ευγενής που δέχτηκε την πρόσκλησή μας. Την επόμενη μάλιστα μέρα από τη συνεδρίαση της Επιτροπής που υιοθέτησε κάποιες ε, διατάξεις και κάποιες συστάσεις για το θέμα που αφορά την ε, εντόλη που έχει λάβει ο ίδιος, τα θέματα που την απασχολούν, δηλαδή τη διεύρυνση. Ξέρετε πολύ καλά ότι το θέμα αυτό είναι συνεχεία αρμοδιότητας του Συμβουλίου τις επόμενες εβδομάδες θα εξεταστούν αυτές οι συστάσεις από το Συμβούλιο. Όπως όλοι ξέρουμε, όμως, και το Κοινοβούλιο και ιδίω η Επιτροπή μας έχει έναν πολύ σημαντικό ρόλο να παίξει για το θέμα αυτό της διεύρυνση. Η δική μα συνένεση είναι μια εκ των όνου προϋπόθεση για την προσχώρηση νέων μελών. Και ο ρόλος μας δεν είναι καθαρά νομικός. Δεν εδράζεται σε μια νομική βάση, αλλά έχει και, ε, παίζουμε και πολιτικό ρόλο. Γιατί η επικοινωνία με τους πολίτες και τους πολίτες των χωρών μας και των πολιτών των χωρών προς ένταξη είναι μια πολύ βασική πτυχή της διαδικασίας της διεύρυνσης. Επομένως, η διεύρυνση δεν είναι μόνο μια τεχνική διαδικασία, προσαρμογή στα πρότυπα, ε, δεν είναι μόνο θέμα διαχείρισης της κρατικής μηχανής ή τρόπου λειτουργίας της ε, κοινωνίας. Μία ένταξη όταν συμβαίνει σημαίνει και προσαρμογή στο σύστημα αξιών που εκπροσωπεί η Ευρωπαϊκή Ένωση στη δικαιοσύνη της, στη δημοκρατία, ε, στα ανθρώπινα δικαιώματα σε όλο αυτό το πλέγμα, το ευαίσθητο των ε, αξιών, ε, είναι πολύ σημαντική η συμμετοχή των πολιτών. Και εμείς λοιπόν ως εκλεγμένοι εκπρόσωποι των πολιτών πρέπει να παίξουμε πρωταγωνιστικό ρόλο στις σχέσεις με, την, ε, με τους πολίτες μας και με την κοινή γνώμη. Επομένως είναι πολύ σημαντικό το καθήκον της προώθησης και διευκόλυνσης των νέων εντάξεων και αυτή η διαδικασία περνάει και μέσα από το Κοινοβούλιο. Και κυρίως μέσω της δικής μας επιτροπής που έχουμε την ειδική εντολή, που ασχολούμαστε ειδικά με αυτά τα θέματα. Θα θέλαμε λοιπόν να γνωρίσουμε τις συστάσεις και τις σκέψεις του Επιτρόπου για το τι συνέβη στο μεταξύ, για τις διάφορες εξελίξεις που έχουν συμβεί. Και ενώ κάνω αυτά τα εισαγωγικά σχόλια, βλέπω ότι μακραίνει ο κατάλογος των συναδέλφων που έχουν ζητήσει να πάρουν τον λόγο. Ζητώ συγγνώμη ακόμα μια φορά για το ότι θα σας πιέσω λίγο από οργανωτικής απόψεως. Σας λέω λοιπόν εκ των προτέρων ότι δεν έχουμε απεριόριστο χρόνο. Θα πούμε λοιπόν εκ των προτέρων δύο λεπτά στον κάθε ομιλητή. Το λέω από την αρχή και χωρίς ε, περαιτέρω εισαγωγές δίνω το λόγο στον ε, Επίτροπο για να μην του κλέψω και άλλο χρόνο. Ευχαριστώ. Thank you very much, uh, for your kind words of uh, introduction. Ευχαριστώ Πρόεδρε για τα ευγενικά σας λόγια που είπατε σαν εισαγωγή. Μεγάλη μου χαρά σας βλέπω όλους σήμερα εδώ. Καταλαβαίνω ότι εδώ πέρα πρόκειται για την ε, αίθουσα των σοσιαλιστών. Α, ήταν, ήταν στο παρελθόν. Σοσιαλδημοκράτες. Καλό είναι να είσαι λίγο παππούς, οπότε χαίρομαι που βρίσκομαι εδώ. Άλλωστε, δεν θα ξεχάσω την υποστήριξη που είχα στην αρχή της διαδρομής μου από τους δημοκράτες. Χθες δε η Επιτροπή ενέκρινε την ετήσια στατική για την στρατηγική διεύρυνση και με την σχετική ανακοίνωση θέλουμε να διατυπώσουμε ότι στα Δυτικά Βαλκάνια σε συγκυρία κρίσης τα πράγματα πάνε καλά και έχουμε κάποιες προκλήσεις που έχουν αντιμετωπίσουν οι χώρες εκείνες αλλά και εμείς στους επόμενου επόμενους μήνες αλλά και χρόνια. Επομένως, είναι πάρα πολύ αυτό σήμερα τα λέμε εδώ σε σχέση με αυτές τις εκθέσεις και πρόκειται για την τελευταία δέσμη θεμάτων διεύρυνσης υπό την ε, τρέχουσα πρώτη Επιτροπή Μπαρός. Σας ευχαριστώ όλους για την ε, εξαιρετική συνεργασία. Κατά το παρελθόν, μια από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ανέκαθεν είχε σημαντικό ρόλο για την διαμόρφωση της πολιτικής ε, διεύρυνσης, ειδικότερα και για την Νοτιοανατολική Ευρώπη, με ψηφίσματα και εκθέσεις. ήταν ε, παράδειγμα προς μίμηση και πιο συγκεκριμένα δική σας επιτροπή ήταν ένας πολύτιμος συνεργάτης σε δύσκολες στιγμές και ελπίζω ότι αυτή η συνεργασία μας θα, συνεργαστεί και στο, θα συνεχιστεί και στο μέλλον. Κυρίες και κύριοι, προσπαθήσαμε την ε, προηγούμενη πενταετία να βρούμε την ε, λεπτή ισορροπία. Απ' τη μια να σταθεροποιήσουμε, να ενδυναμώσουμε και να είμαστε ταυτόχρονα συνεπείς στις ε, δεσμεύσεις μας για ευημερία, δημοκρατία, ελευθερία. Γιατί θα πρέπει από την άλλη μεριά κανείς να εξασφαλίσει την δυνατότητα ένταξης και ενσωμάτωσης. Και έτσι προχωρήσαμε με πάρα πολύ προσεκτική διαχείριση για να δούμε πώς η διαδρομή προς την Ευρωπαϊκή Ένωση θα είναι πιο αποδοτική για τις ενδιαφερόμενες χώρες. Οπότε τώρα θέλω να σταθώ σε κάποια παραδείγματα, δύο συγκεκριμένα, για όσα σας είπα πρώτα-πρώτα. Τώρα μπορούμε να συστήσουμε την έναξη των διαπραγματεύσεων με την πρώην Ιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας. Μας έχει πείσει ότι έχει προοδεύσει αυτή η χώρα και επίσης ότι ξεκίνησε κάποιες κρίσιμες μεταρρυθμίσεις στην δικαιοσύνη, την αστυνομία, την δημόσια διοίκηση και την εφαρμογή του, της συμφωνίας πλαίσιο για την προστασία των μειονοτήτων. Και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θεωρεί ότι επομένω πληρεί η χώρα αυτή τα κριτήρια που έταξε η συνάντηση της Κοπενχάγης. Οπότε θα πρέπει τώρα να δούμε πώς θα καλυφθούν οι βασικές προτεραιότητε και κατά πόσον πληρούνται τα πολιτικά κριτήρια, ούτω ώστε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να φτάσει σήμερα στο να προτείνει την άρχιση των διαπραγματεύσεων. Φαντάζομαι ότι όλα αυτά είναι πολύ σημαντική ενθάρρυνση για τα Σκόπια, ούτως ώστε να ξεκινήσουν, να ολοκληρώσουν τις συνομιλίες για το θέμα της ονομασίας. Χθε. είπαμε πίσω ότι θα πρέπει να, έχουν, να υπάρχουν καλές γειτονικέ σχέσεις και να βρεθεί όσον αφορά την ονομασία μια αμοιβή αποδεκτή λύση υπό την αιγίδα του ΟΗΕ. Είναι πολύ σημαντικό αυτό το θέμα και τώρα. Αυτό θα πρέπει να διεκπαιρεωθεί γιατί είναι πάρα πολύ επίγον εν ώψη του ευρωπαϊκού μέλλοντος της χώρας. Φαντάζομαι ότι αυτό το μήνυμα το οποίο στείλαμε έχει ληφθεί από τα Σκόπια. Δεύτερον, η απορρίθμιση στα Δυτικά Βαλκάνια έχει προχωρήσει φέτος και θα συνεχιστεί αυτή η πορεία και του χρόνου συζητούνται οι προτάσεις και όσον αφορά τις θεωρίες διαβατηρίων για πρώην Ιουγκοσλαβική Δημοκρατία Μακεδονίας, Μαυροβούνια και Σερβία και την άρση των σχετικών περιορισμών από πρώτης πρώτη του επόμενου έτους. Μια που πλήρωνται όλες οι σχετικές προϋποθέσεις, Φερρυπίν, τα μοντέρνα διαβατήρια, τα βιομετρικά και κάποια μέτρα για τις ε, μεθορίους, τα σύνορα, ούτω ώστε να υπάρχει άριστο προορισμό σε αφορά τις ε, θεωρήσεις και να θεωρηθεί ότι για τους Ευρωπαίους πολίτες υπάρχει ασφάλεια. Ξέρω ότι θα περιμένατε, και εγώ ίσως θα το ήθελα, να έχουμε πιο πολλά στοιχεία να, έχουμε πιο, να είναι πιο σφαιρική αυτή η έκθεση, αλλά για Βοσνία, για Ζεγοβίνη και Αλβανία έχουμε βάλει κάποιε αυστηρέ προποθέσει όσον αφορά τι θεωρήσει, ούτω ώστε να μπορέσουμε να πείσουμε του υπουργού εσωτερικών και θα υποβάλουμε κάποιε προτάσει για Βοσνία και Αλβανία κατά το πρώτο εξάμεινο του επόμενου έτου. ανάλογα με το τι έχουν κάνει αυτές οι χώρες για τις προποθέσεις που έχει τάξει ο της πορείας σχετικός. Πολύ σημαντικά αυτά τα ζητήματα για τους κατοίκους των χωρών και ιδίω για τους ε, σπουδαστές και φοιτητές οπότε και βλέπετε πόσο αυτές μας οι προτάσεις ωφελούν χειροπιαστά του κατοίκου των χωρών αυτών. Και βλέπουμε έναν κάποιο εξευρωπαϊσμό των κοινωνιών εκείνων και αυτό είναι άλλωστε ο βασικό στόχος. Σκεφτείτε τι γινόταν πριν από μία πενταετία. Ούτε καν μπορούσε να διανοηθεί κανεί ότι θα έχουμε διευκολύνσει πόσο μάλλον κατάργηση τη θεώρηση διαβατηρίου. Αυτά είναι τα, τα ωφελήματα από την διεύρυνση που προκύπτουν για τις χώρες εκείνες. Η ευρωπαϊκή προοπτική για Δυτικά Βαλκάνια αλλά και Τουρκία ήταν ε, ένας παράγων σταθερότητας για το δημοκρατικό μετασχηματισμό. Να δούμε τώρα τι χώρε χώρες, λίγο να όχι, όχι όλες, ε, ίσως ε, να το συζητήσουμε έτσι σαν, ένα διάλογο το τι γίνεται. Η Κροατία θα είναι μάλλον 28η χώρα που θα μπει στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Βρίσκεται κοντά στη γραμμή του τερματισμού μετά από μια πορεία τετραετή όπου είχαμε εντατικές επαφές για την διεύρυνση. Θα πρέπει η χώρα να συνεχίσει τις προσπαθειές της, τις μεταρρυθμιστικές, ιδίως για δικαιοσύνη, κατά πολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος, διαφθοράς και να συνεργαστεί με το Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης πριν θεωρήσουμε ότι έχουν ολοκληρωθεί οι διαπραγματεύσεις. όχι τώρα μια καινούργια όθηση αυτή η υπόθεση γιατί η Κροατία πληρεί τις σχετικές προϋποθέσεις για την προσχώρηση οπότε οι διαπραγματεύσει κατά την επόμενη χρονιά θα ολοκληρωθούν. Για τα υπόλοιπα Δυτικά Βαλκάνια επίσης γίναμε μάρτυρες μιας ε, σταθερής ε, αλλά βέβαια άνηση ε, πορείας σταθεροποίηση πέρσι και είχαμε κάποιες συμφωνίες ελευθερών εμπορίου για τις υπόλοιπες χώρες της ε, περιοχής, ε, πρώην Ιουγκοσλαβία, Δημοκρατία Μακεδονία, Αλβανία, Βοσνία, Σερβία, αλλά και Κόσοβο. Οπότε, με δεδομένη αυτή τη σταθεροποίηση, θα πρέπει να εξασφαλιστεί η ειρήνη και να είμαστε σίγουροι ότι θα συνεχιστεί αυτή η κατάσταση. Οπότε και εμείς θα πρέπει να συνεχίσουμε αυτό το οποίο θα μπορούσα να το ονομάσω ω πολιτική ναρκαλίευση στα Δυτικά Βαρκάλια, ούτω ώστε να αποφύγουμε τα πισωγυρίσματα. Επίσης με μαρτύρε κάποιων επιτυχιών, όπως αυτή η συμφωνία για την ε, συνοριακή διαφορά μεταξύ Σλοβενίας και Κροατίας. Ε, γίναμε οι διαμεσολαβητέ ως Ευρωπαϊκή Ένωση και κατά αυτόν τον τρόπο δόθηκε και νέα όθηση στις προσπάθειες της ε, προσχώρηση της Ευρωπαϊκή Ένωση μετά από το φρενάρισμα που είχε γίνει για σχεδόν μια χρονιά. Αλλά πρέπει να ξανασυνεχίσουμε την προσπάθεια. Υπάρχει ένα σημείο το οποίο συζητείται αυτή τη στιγμή με τις διαπραγματευτικές μας ομάδες στο Σαράγεβο, στο Μούσταρ. Αναφέρομαι βέβαια στη Βοσνία Ερσεγοβίνη, που κινδυνεύει να μείνει πίσω και να καθυστερήσει σε σχέση με τι υπόλοιπε χώρε τη περιοχή. Την περασμένη εβδομάδα, λοιπόν, μαζί με τον Πρωθυπουργό Καρλ Μπίλτ ε, των Υπουργών Εξωτερικών και τον κύριο ε, Στάιμπερκ τον Αμερικανό, ε, συναντηθήκαμε επί δύο μέρες με ηγέτες κομμάτων της Βοσνίας Τσεγοβίνης για να ξεπεράσουμε το αδιέξοδο που κρατάει πίσω τη χώρα αυτή τους τελευταίους μήνες. Θα ξαναπάμε την επόμενη εβδομάδα Όπως σας είπα, οι διαπραγματευτικές μας ομάδες ε, συνεχίζουν τις συνομιλίες με τους ηγέτες της χώρας. Έχουμε προσφέρει ένα πακέτο μέτρων στη χώρα που συμπεριλαμβάνει και κάποιες συνταγματικές μεταρρυθμίσεις που θα τους βοηθήσουν για να ξεκινήσουν την ε, ενταξιακή πορεία προς την Ευρωπαϊκή Ένωση και στο ΝΑΤΟ. Γιατί το κάνουμε αυτό. Γιατί θέλουμε η Βοσνία και η Ζεγοβίνη να είναι μια αξιόπιστη υποψήφια χώρα για την ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στο ΝΑΤΟ. Πρέπει να ξεκαθαρίσουμε ότι μια υποψηφιότητα για την ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση από τη Βοσνία και την Ερζεγοβίνη μπορεί να αρχίσει να εξετάζεται μόνο όταν το θέμα του OHR ε, έχει κλείσει. Δεν μπορεί ένα σχεδόν προτεκτοράτο να ξεκινήσει την ε, ένταξή της στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Επομένως, οι ηγέτες και τελικά ο λαός της Βοσνίας Ερζεγοβίνης πρέπει να αποφασίσει εάν η χώρα θέλει να παραμείνει μόνιμα πίσω από τους υπόλοιπους σε κάποια μορφή ενταξιακής έτσι, σχέσης με την Ευρωπαϊκή Ένωση μια σχέση σύνδεση ή να ξεκινήσει την ενταξιακή της πορεία ε, με, με όλες τις προϋποθέσεις όμως που απορρέουν. Ελπίζω ότι οι πολίτες της Βοσνίας Ερσεγοβίνης και οι ηγέτες για το καλό της χώρας και της περιοχής συνολικά των Δυτικών Βαλκανίων θα προσπαθήσουν να πετύχουν την ένταξη της, της χώρας τους στην ε, Ευρωπαϊκή Ένωση και στο ΝΑΤΟ. Σε αυτές τις δύσκολες στιγμές οικονομικής κρίσης, οι αιτήσει ε, για την ένταξη του Μαυροβουνίου και της Αλβανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση δείχνουν την ε, έλξη που ασκεί η Ευρωπαϊκή Ένωση στις χώρες αυτές και στο πόσο πιστεύουν ότι προωθούμε τη σταθερότητα, την ασφάλεια και την ευημερία. Η αίτηση της Ισλανδίας ε, για την ένταξή της δίνει επίσης μια νέα διάσταση στην ατζέντα της διεύρυνσης, όχι μόνο γεωγραφικός πώς και στρατηγικός πώς, αλλά και γιατί ε, μόνο έτσι αυτή η χώρα θα εξασφαλίσει την ε, οικονομική σταθερότητα, μια χώρα που έχει πάρα πολύ πληγή από την οικονομική κρίση. Πριν καταλήξω, θα ήθελα να τονίσω κάποιες βασικές προκλήσεις που μας περιμένουν στην περιοχή. Πρέπει να ξεκινήσω με το κράτος δικαίου, που είναι μια θεμελιώδης ευρωπαϊκή αξία και που είναι μια μεγάλη πρόκληση στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Μιλάω ειδικά για τη μεταρρύθμιση της δικαιοσύνης και την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος. Γίνονται πάρα πολλά στον τομέα και η Κομισιόν χρησιμοποιεί όλα τα κοινοτικά μέσα για να βοηθήσει αυτές τις χώρες στις προσπάθειές τους να αντιμετωπίσουν τη διαφθορά και το έγκλημα. Είναι μια μεγάλη προτεραιότητα και έχουμε διδαχθεί πολλά από τις προηγούμενες ε, προσπάθειες, ε, τους προηγούμενους γύρους Δυστυχώς, η ελευθερία έκφρασης και η ελευθερία των μέσων ενημέρωσης ε, παραμένουν ε, πρόβλημα σε πολλές χώρες της περιοχής. Και αυτό θα πρέπει να αντιμετωπιστεί με τρόπο κατεπήγοντα και με πιστικό τρόπο από τις ενδιαφερόμενες χώρες. Παραδείγματο χάρη, ήμασταν ξεκάθαροι απέναντι στην Τουρκία ότι η ελευθερία σκέψης, λόγου και τύπου είναι θεμελιώδες, θεμελιώδεις αξίες, οποιαδήποτε ανοιχτή και δημοκρατική κοινωνία και είναι εκ των όνων καν προϋπόθεση για την ένταξή της στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Το ίδιο ισχύει για τις θρησκευτικέ ε, ελευθερίες, τα δικαιώματα των γυναικών και τα δικαιώματα των μειονοτήτων. Καθώς και τα δικαιώματα των συνδικάτων βέβαια. Τώρα, στο ευρύτερο στρατηγικό πλαίσιο, η Τουρκία παίζει ένα σημαντικό ρόλο στην ε, περιφερειακή ασφάλεια, παραδείγματο χάρη στην ε, Μέση Ανατολή, στον Νότιο Κάφκασο, εξασφαλίζει την ενεργειακή ασφάλεια και παίζει σημαντικό ρόλο στην προώθηση του διαλόγου μεταξύ πολιτισμών. Αυτοί είναι βασικοί λόγοι για τους οποίους ξεκινήσαμε στην, ε, με την ενταξιακή διαδικασία της ε, Τουρκίας. Επίσης καλωσορίζω την εξομάλυνση των σχέσεων με την Αρμενία που είναι μια ιστορική στιγμή, ένα ιστορικό βήμα, κάτι που καλωσορίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί θεωρείται σημαντική συνεισφορά σταθερότητα και στην ειρήνη στην περιοχή. Επίσης, καλωσορίζω το δημοκρατικό άνοιγμα ε, για την επίλυση του Κουρδικού με ευρεία διαβούλευση και συγκεκριμένα μέτρα. Περιμένουμε ότι η Τουρκία θα εξασφαλίσει την πλήρη εφαρμογή του επιπρόσθετου πρωτοκόλλου της Συμφωνίας Σύνδεσης που ονομάζεται Συμφωνία της Άγκυρας του 1963 και περιμένουμε ότι η Τουρκία θα κάνει πρόοδο για την ε, εξομάλυση των σχέσεων με την Δημοκρατία της Κύπρου. Ζητούμε από τους ηγέτες των δύο κοινοτήτων στην Κύπρο να ολοκληρώσουν επιτυχώς τις ε, συνομιλίες διευθέτησης και ζητούμε από την Τουρκία να συνεισφέρει με συγκεκριμένο τρόπο σε μια επίλυση του Κυπριακού, ευρύ επίλυση. Κάποια άλλα μακροπρόθεσμα προβλήματα στην περιοχή είναι διμερεί θέματα. Οι διμερείς ε, διενέξεις θα πρέπει να επιληθούν από τα ενδιαφερόμενα μέλη και δεν θα πρέπει να δημιουργήσουν προσκόμματα στην ε, ενταξιακή διαδικασία. Η περιφερειακή συνεργασία στην Νοτιοανατολική Ευρώπη έχει βελτιωθεί το 2009 και ήταν μία από τις βασικές προτεραιότητές μας αυτές, αυτή. Οι χώρες στην περιοχή ασχολούνται όλο και περισσότερο με την διαδικασία της ε, περιφερειακής ε, συνεργασίας σε πολιτικό επίπεδο, στα πλαίσια του Περιφερειακού Συμβουλίου Συνεργασίας ή οικονομική συνεργασία στα πλαίσια της ε, Συμφωνίας Ελευθέρου Εμπορίου. Όμως η αποτελεσματικότητα των περιφερειακών δομών θα πρέπει να βελτιωθεί και οι διαφωνίες για το κοσφοπέδιο δεν θα πρέπει να αποτελέσουν πρόσχομα στην περιφερειακή συνεργασία. Κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, αγαπητοί βουλευτές, θα ήθελα να καταλήξω τονίζοντας ότι η πολιτική διεύρυνσης παραμένει στρατηγικό συμφέρον της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μας βοηθάει να προβάλλουμε την σημασία και επιρροή της Ευρωπαϊκής Ένωσης πέρα από τα σημερινά μας σύνορα και χρησιμεύει ως πόλος σταθερότητας σε αυτές τις δύσκολες στιγμές. Η πολιτική μας για τη σταθερότητα μερικές φορές συμπίπτει με την πολιτική διεύρυνσης. Είχε και έχει σοβαρότητες ε, επιπτώσεις ε, στην εξωτερική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στον ε, παγκόσμιο της ρόλο. Με άλλα λόγια, η αξιοπιστία μας ως ε, παγκόσμιο τέρου βασίζεται σε μεγάλο βαθμό στην ικανότητά μας να διαμορφώσουμε τη δική μας άμεση γειτονία μέσω της πολιτικής γειτονίας και μέσω της διεύρυνσης. Η ικανότητα μετασχηματισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι μεγαλύτερη στην νότια και ανατολική γειτονιά μας, όπου ο τρόπος ζωής που βασίζεται στη δημοκρατία και στις θεμελιώδεις ελευθερίες δίνουν ελπίδα και οδηγούν στις μεταρρυθμίσεις. Εκεί λοιπόν μπορούμε να παίξουμε κάποια, κάποιο ρόλο και να κάνουμε τη διαφορά. Πέρα από τα τεχνικά στοιχεία της έκθεσης πρόοδου, αυτή είναι η ιστορία που μας ενδιαφέρει. Αυτή είναι η έλξη που ασκούμε στην περιοχή. Επομένως, ε, η Νοτιοανατολική Ευρώπη, η Ανατολική Γειτονία και η Ένωση για τη Μεσόγειο θα πρέπει να παραμείνουν βασικέ προτεραιότητε τη Ευρωπαϊκή Ένωση, καθώ και η ειρήνη στη Μέση Ανατολή, η σχέση με το Ιράν, η σταθερότητα στο Νότιο Κάφκασο, η ενεργειακή ασφάλεια, η καταπολέμηση τη δημοκρατίας, όλα αυτά είναι θέματα τα οποία δεν μπορούμε να αντιμετωπίσουμε ούτε να επιλύσουμε μόνοι μας. Χρειαζόμαστε τέρου. και χρειαζόμαστε και τους εταίρους της νοτιοανατολικής ε, Ευρώπης να μας βοηθήσουν σε αυτήν την προσπάθεια. Αγαπητοί φίλοι, μόνο με αυτόν τον τρόπο μπορούμε να παίξουμε το ρόλο μας για την ειρήνη, την ε, σταθερότητα, τη δημοκρατία. Αυτές είναι βασικές αξίες. Νομίζω ότι αυτή είναι η βασική μας αποστολή και σε αυτή τη διαδικασία το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα μας βοηθήσει πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ αγαπητέ Επίτροπε. Η παρέμβασή σας ήταν πάρα πολύ ευρεία, πλήρης και πολύ ενδιαφέρουσα. Ήταν τόσο ενδιαφέρουσα που 26 συνάδελφοι μου ζητούν το λόγο. Δυστυχώς θα σας κλέψω κι άλλο χρόνο, θα σας περιορίσω κι άλλο το χρόνο. Από δύο λεφτά, ενάμιση. Θα δώσω καταρχάς ε, πρώτα το λόγο στους ε, εισηγητές. Ο πρώτος που έχει το λόγο είναι η κυρία Πακ. Ehm, Συγητρία και διακόπτη η κυρία Πακ όμως. Ευχαριστώ. Δεν θα μιλήσω όμως μόνο για τη Βοσνία. Κύριε Επίτροπε, σας ευχαριστώ για τις εισαγωγικές σας παρατηρήσεις. Αναφερθήκατε στη Μακεδονία. Διερωτηθήκατε αν τα Σκόπια αντελήφθησαν το μήνυμα. Εγώ θέλω να ρωτήσω αν και η Αθήνα κατάλαβε το μήνυμα. Γιατί μόνο τα Σκόπια, μόνο η Μακεδονία, μόνοι τους δεν μπορούν να στρέψουν την πορεία προς ε, ε, ένα, ε, να στραφούν προς μια ορθή πορεία. Πρέπει και η Ελλάδα να συμβάλλει. Ελπίζω ότι το κατανοεί αυτό η Ελλάδα. Το θέμα της ε, προξενικής θεώρησης θα μας απασχολήσει και τις επόμενες εβδομάδες. Νομίζω ότι ήταν λάθος να προβεί σε αυτές τις διαφοροποιήσεις η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τον Ιούνιο. Το μόνο που μπορεί να γίνει τώρα είναι να πει καθαρά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι του χρόνου θα μπορέσει να συμβάλλει. Το θέμα του Κωσόβου εν προκειμένου είναι σημαντικό. Πρέπει να προσφέρουμε κάθε δυνατή βοήθεια στο Κόσοβο ώστε να μην γίνει εκεί μια πραγματική μαύρη τρύπα. Για την Κροατία δεν χρειάζεται να πω τίποτε, γιατί βρίσκεται σε καλό δρόμο. Για την Βοσνία Ριζεγοβίνη νομίζω ότι αυτή η ιστορία ε, προχώρησε πάρα πολύ γρήγορα και χωρίς καλή προετοιμασία και ίσως είναι καταδικασμένη σε αποτυχία. Εάν δεν βασιστούμε σε κάτι το οποίο ήδη έχει γίνει αντικείμενο διαπραγμάτευση εκεί. Ήδη υπάρχει μια συμφωνία. Ίσως λοιπόν μπορεί να στραφεί προς κάποια καλύτερη κατεύθυνση. Με κατέπληξε το ότι δεν αναφερθήκατε καθόλου στην Αλβανία, μια χώρα η οποία έχει κάνει πρόοδους, έχει τώρα μια καλή και σταθερή κυβέρνηση και επαναλαμβάνω με αυτό με κατέπληξε. Ε, νομίζω ότι ε, σεβάστηκα το χρόνο μου. Μην κάνετε παραπάνω από δύο ερωτήσεις. Αυτή είναι η ε, παρακλησή μου προς όλους. Όμεν Ρόιτεν, Τουρκία. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η κυρία Πακ ήδη κάλυψε όλα τα Βαλκάνια. Άρα εγώ θα αναφερθώ μονάχα στην Τουρκία. Διεπίστωσα ότι ο Επίτροπος ε, κ. Ρέινς, ό,τι αφορά την Τουρκία, ήταν επικριτικός. Σημείωσα επίσης ότι είπε ότι σε κάθε διεύρυνση πρέπει να τονίζεται η ανάγκη να υπάρχει κράτος δικαίου. Η Τουρκία βέβαια πρέπει να το πράξει αυτό, δηλαδή να θεσπίσει πραγματικό κράτο δικαίου και προ το δικό τη συμφέρον, το ίδιο συμφέρον. Διότι αυτό αποτελεί και την βασική προϋπόθεση για κάθε εξέλιξη. Έχω τώρα τρεις ερωτήσεις. Πρώτη, είπε ο κύριος Επίτροπος σήμερα ότι αναμένει να γίνει ε, σεβαστό το πρόσθετο πρωτόκολλο. Έτσι είπε, αλλά στην έκθεση δεν λέει τίποτα τέτοιο. Τι ισχύει τώρα, τα λεγόμενα ή τα γραπτά. Δεύτερο, η μεταρρύθμιση της δικαιοσύνης. Στην έκθεσή σας λέτε ότι έχει γίνει μια αρχή και ότι αν δεν γίνουν αρκετά πράγματα τότε δεν μπορεί να προχωρήσει η υπόθεση με την Τουρκία. Αυτά ήθελα να πω. Παρακαλώ, να σεβαστούμε όλοι τον χρόνο. Τάλερ. Ε, σας ευχαριστώ κύριε Επίτροπε για το έργο σας, για το θάρρος σας ειδικότερα για τη Μακεδονία που προτείνεται να αρχίσουν διαπραγματεύσεις μετά από μια τετραετία χθες στο κέντρο των Σκοπίων έγινε πανηγύρι και μπορεί να δει κανείς τι σημασία αποδίδει όχι μόνο η κυβέρνηση των Σκοπίων αλλά και ο λαός της Μακεδονίας στην διαδικασία αυτή. Τώρα, ποιε πιστεύετε ότι είναι οι πιθανότητε να υποστηρίξει το Συμβούλιο την απόφαση αυτή, Βλέπετε να υπάρχει ένα λεγόμενο παράθυρο ευκαιρία μετά από τι πρόσφατε ελληνικέ εκλογέ. Βλέπουμε τώρα τον κύριο Παπανδρέου που επανήλθε στο αξίωμα του Πρωθυπουργού και ο οποίο είναι ο αρχιτέκτονα τη ατζέντα Θεσσαλονίκη του 2003. Θυμίζω και τον λόγο του Πρωθυπουργού Γκρουέλσκι πριν από λίγες μέρες, γιατί φάνηκε πολύ θετικό στον λόγο του, λόγο που εκφωνήθηκε για μια εθνική γιορτή της 11ης Οκτωβρίου και τόνισε ότι είναι ανάγκη να υπάρξει κοινή συμφωνία για τα διμερεί προβλήματα περιλαμβανομένης και της ονομασίας. Βλέπετε να υπάρχει κάποια πρόοδο όπω είδατε και στην περίπτωση τη Κροατία και τη Σλοβενίας στην ε, σύγκρουση αυτή δηλαδή. Σας ευχαριστώ που σεβαστήκατε και το χρόνο σα, κύριε Τάλιν. Ε, ο εισηγητή για τη Σερβία, ο κύριος Κάτσιν, 1,5 λεπτό. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Κύριε Επίτροπε, θα ήθελα να σας συγχαρώ για όλα όσα πετύχατε αυτό το διάστημα. Μόνο για τη Βοσνία Ζεγοβίνη διακόπτει ο, ο Επίτροπος. Θα ξεκινήσω με τη Σερβία και θα μιλήσω για όλα τα Δυτικά Βαλκάνια και για την Τουρκία. Θα ήθελα να τονίσω ότι είναι εξαιρετικά σημαντικό το γεγονός ότι είσαστε αισιόδοξο. Το γεγονός ότι δημιουργείται πάντα ε, μια θετική ατμόσφαιρα. Γιατί η θετική ατμόσφαιρα είναι μια προϋπόθεση όχι μόνο για τα Δυτικά Βαλκάνια, αλλά για την πολυμερή προσέγγιση που θέλουμε να προωθήσουμε σε όλο τον πλανήτη. Θα ήθελα καταρχάς να σας συγχαρώ εσάς προσωπικά για την αγγελία του σχεδίου να συμπεριλάβατε και το κοσυφοπαίδιο στο καθεστώς απελευθέρωσης των θεωρήσεων. Είναι μια μεγάλη στιγμή για τα Δυτικά Βαλκάνια και για τη Σερβία. Θα ήθελα λοιπόν να σας ρωτήσω αν υπάρχει κάποιο χρονοδιάγραμμα για να, ξεκινήσουν, να ξεκινήσει αυτή η διαδικασία. Και όχι απλώς να ξεκινήσει, αλλά να εφαρμοστεί κιόλα. Ε, με προκαλέσατε τώρα για τη Βοσνία Ζεγοβίνη, έτσι. Ε, έρχομαι από τον Μπουτιμίρ και νομίζω ότι η λειτουργία της ε, βοσνιακής κυβέρνησης ε, ε, γύρει κάποια θέματα, υπάρχουν κάποιες προκλήσεις. Μιλήσατε για διμερεί θέματα, για την έκτηση προόδου για την Κροατία και το θέμα των συνόρων. Δεν υπάρχει πρόοδος στο θέμα των συνόρων στη Βοσνία-Ερσεγοβίνη. Χωρίς καλή διακυβέρνηση εκεί στη Βοσνία-Ερσεγοβίνη υπάρχει περίπτωση να δημιουργηθεί κάποιο κάποια πρόοδο στο θέμα των συνόρων. Ευχαριστώ. Κύριος Λούνατσεκ, κυρία Λούνατσεκ, που είναι η για το κοσφοπέδιο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε. Αρχίζοντας, θα ήθελα να πω, όπως είπαν και ορισμένοι άλλοι, ότι είμαι ιδιαίτερα ικανοποιημένη διότι επανεπιβεβαιώσατε την ευρωπαϊκή προοπτική όλων των χωρών των Δυτικών Βαλκανίων διότι γνωρίζω ότι ορισμένες χώρες μέλη δεν το βλέπουν με τον ίδιο τρόπο. Γι' αυτό το λόγο και είμαι ιδιαίτερα ικανοποιημένη. Ω εισηγήτρια για το Κόσοβο είμαι άλλωστε ακόμη πιο ικανοποιημένη διότι περιλάβατε και το Κόσοβο στην προοπτική ε, των νέων ρυθμίσεων για τις προξενικές θεωρήσεις. Οι πολίτες του Κόσοβου το περιμένουν αυτό. Αυτό το στοιχείο που λείπει τώρα είναι να μας πείτε πότε θα αρχίσει το διάλογο αυτό. Το άλλο είναι οι πληθυσμοί Ρώμα στο Κόσοβο. Στην έκθεσή σας και σωστά αναφέρετε ότι υπάρχουν ακόμη πολλές προκλήσεις. Ξέρουμε τώρα ότι γίνονται διαπραγματεύσεις για συμφωνίες επανεισδοχής με όλες αυτές τις χώρες. Ασκείται πίεση στις χώρες μέλη να μην στέλνουν τους Ρώμα πίσω στο Κόσοβο όπου η κατάστασή τους δεν είναι ξεκάθαρη και προκαλούνται σημαντικά προβλήματα. Νομίζω ότι οι χώρες μέλη πρέπει και αυτές να δουν ακριβώς πού θα ε, στείλουν πίσω τους Ρώμα. Τέλος, για την Τουρκία, αν και θα τα πει ο συναδελφός μου περισσότερα, ευρωπαϊκές προδιαγραφές, για παράδειγμα και για υδροελεκτρικά εργοστάσια όπως το φράγμα του Λίσο. Ευχαριστώ την κυρία Λούνατσεκ. Κούκαν, πρόεδρος της αντιπροσωπείας για τις χώρες των, της Νοτιοανατολικής Ευρώπης. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε και ευχαριστούμε και τον Επίτροπο Ρεν για τόσο μας εξέθεσε. Είπαν οι προηγούμενοι αγορητές ότι υπάρχουν κάποια καλά νέα για την ε, περιοχή αυτήν και για τις χώρες ε, πιο συγκεκριμένα και ο κύριος Επίτροπος επίσης ε, σύντομα μας είπε ότι θα ήταν σωστό το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να εκμεταλλευτεί την ευκαιρία αυτής της ε, συγκυρίας ούτω ώστε να ενδυναμώσει και την παρουσία του και σας ρωτώ πώς θα πρέπει να γίνει αυτή η συνεργασία θα πρέπει να γίνει έτσι ούτω ώστε να υπάρχει ε, κάποια απτή συμβολή στην διαδικασία αυτή. Κύριε Τάνοκ, είστε εισηγητής για το Μαυροβούνιο. Ε, σας δίνω κατ' το λόγο γιατί ζητήσατε κατόπιν εορτή το λόγο. Εν πάση περιπτώσει, τον έχετε. Δεν θα με ακριβώς. Διάβασα την έκθεση πρόοδου του Μαυροβουνίου και από ό,τι φαίνεται υπάρχει πρόοδος σε όλους τους ε, τομείς, κάποια πρόοδος και έχουμε περί, περί τα 2.000 γραπτέ ερωτήσει που απίθυνε προ την κυβέρνηση και Κομισιόν και βέβαια για μια μικρή χώρα που δεν έχει σπουδαία διοίκηση πρέπει να πούμε ήταν Ηράκλειε οι προσπάθειε που κατέβαλαν τόσο ώστε να μπορέσουν να ανταποκριθούν σε αυτέ τι ε, απαιτήσει για, για την υποψηφιότητα και καταπολεμούν όσο μπορούν την διαφθορά, το ερωμένο έγκλημα και ένα από τα προβλήματα που ακόμη εκκρεμούν είναι το, το, η, η προθεσμία όσον αφορά την ε, συμφωνία ε, σταθερότητας και σύνδεσης που ακόμα δεν έχει κυρωθεί από κάποιες χώρες και το Ηνωμένο Βασίλειο ακόμα δεν έχουν κυρώσει αυτή τη σχετική συμφωνία. Επομένως, αυτό είναι πρόβλημα και θα πρέπει στα εθνικά κοινοβούλια να, να, να, αποκτήσει το θέμα προτεραιότητα και να αρθούν τα σχετικά προβλήματα στο Συμβούλιο. Η οικονομία του Μαυρομνίου φύγει από την κρίση βέβαια. Ε, κυρίως ε, ο τουριστικός τομέας ε, ανθεί, έχει ένα-δύο εργοστάσια σημαντικά, βιομηχανίες. και προς να καταφέρουν. Επίσης ε, το θέμα με τα βιομετρικά διαβατήρια ήταν σημαντικό και για την άρση της θεώρησης διαβατήριων. Ευχαριστώ κύριε Τάνο. Κλείνουμε με αυτή την παρέμβαση την πρώτη ομάδα ερωτήσεων και τώρα το λόγο έχει ο Επίτροπος να απαντήσει. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ και όλους τους υπεύθυνους σε αυτές τις εύστοχες ερωτήσεις. Ξεκινώ με τις ερωτήσεις της Doris Πακ και της για τα Σκόπια. Χθες, αυτό το οποίο προτείναμε, είχε δύο στόχους. Δηλαδή αυτή η σύσταση του να αρχίσουν οι ενταξιακές διαπραγματεύσεις με την πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας. Θα πρέπει... Είναι δυτή η ενθάρρυνση αυτή που γίνεται και θέλουμε να τους ενθαρρύνουμε τόσο ώστε να συνεχίσουν τις μεταρρυθμίσεις τους όσον αφορά το δίκαιο, όσον αφορά την δημοκρατία και να πετύχουν κάποιες συγκεκριμένες επιδόσεις και αποτελέσματα, αλλά ταυτόχρονα τους ενθαρρύνουμε σημαντικά ούτως ώστε να ξεκινήσουν κάποιες σοβαρές διαπραγματεύσεις με θετικό πνεύμα οπότε και το θέμα αυτό να τακτοποιηθεί. Είμαι σε τακτικές επαφές με τον κύριο Νίμιτς που είναι ο διαμεσολαβητής του ΟΗΕ για το θέμα της ονομασίας. Εδώ και 15 χρόνια ασχολείται με αυτό και κάνει μια θαυμάσια δουλειά. Παρότι δεν έχουν επιτευχθεί ακόμη αποτελέσματα. Αυτό δεν οφείλεται στη δική του έλλειψη προσπάθειας. Αντίθετα, τώρα έχει αρκετή αισιοδοξία και στις αρχές του φθινοπόρου μάλιστα η αισιοδοξία αυτή ήταν πολύ πιο έντονη. Θεωρεί λοιπόν όταν αναλάβουν οι νέες ε, κυβερνήσεις ε, με μια νέα εντολή, πραγματικά θα δημιουργηθεί ένα νέο παράθυρο ευκαιρίας για να, δημιουργηθεί αυτό το, λυθεί αυτό το θέμα που μας ταλανίσει εδώ και 18 χρόνια. Γνωρίζω ότι στο Συμβούλιο χρειαζόμαστε ομοφωνία για να ξεκινήσουν διαπραγματεύσεις ένταξης με οποιαδήποτε χώρα. Το ξέρουμε αυτό. Και Πιστεύουμε ότι με την πρότασή μας θα εξασφαλίσουμε και συνθήκες καλής γειτονίας ε, και για αυτές ε, η επίλυση του θέματος ονομασίας είναι βασική προϋπόθεση. Νομίζω ότι αυτό το μήνυμα έχει περάσει και στα Σκόπια και παντού. Για το θέμα των θεωρήσεων. Συμφωνώ μαζί σας ότι αυτή τη στιγμή οι χώρες ε, σεβαστούν τις προϋποθέσεις η Βοσνία Σεγοβίνη και η Αλβανία δηλαδή, μπορούμε να συστήσουμε την απελευθέρωση από το καθεστώς των θεωρήσεων για τους πολίτες τους. Φυσικά αυτό το θέμα εμπίπτει στον Επίτροπο που ασχολείται με θέματα δικαιοσύνης, ασφάλειας και ελευθερίας. Είναι θέμα δηλαδή του Ζακ Μπαρό. Ε, έχουμε συνεργαστεί θαυμάσια ε, μαζί για το θέμα των θεωρήσεων για τα Δυτικά Βαλκάνια. Και επίσης ε, είμαι ευγνώμων και για την υποστήριξη που μου έδωσε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για αυτό το θέμα. Και για τις ε, απόψει που έχετε εκφράσει τα τελευταία χρόνια. Οι προσπάθειες που έχει κάνει η Βοσνία Σεγοβίνη δεν μπορούν να χαρακτηριστούν αποτυχία. γίνεται μια σοβαρή προσπάθεια και μάλιστα η προσπάθεια είναι κοινή ε, Ευρωπαϊκής Ένωσης, Ηνωμένων Πολιτειών, σε υψηλότατο επίπεδο, η Προεδρία, το Συμβούλιο, η Κομισιόν από πλευράς Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και ο κ. Στάιμπεργκ, ο Υφυπουργό ε, Εξωτερικών, με την ε, υποστήριξη του Πρόεδρου Ομπάμα και την Υπουργό Εξωτερικών, την Χίλαρη Κλίντον, προσπαθούμε να βοηθήσουμε την Βοσνία Σεγοβίνη στην ενταξιακή της πορεία στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στο ΝΑΤΟ. Το θέμα των Ρώμα θέτουν και το θέμα του κράτους δικαίου στην Τουρκία. Η έκθεσή μου τονίζει ότι πρέπει να επανεκκινήσει η διαδικασία μεταρρύθμισης. Ε, μιλάω για τα δικαιώματα των γυναικών, των μειονοτήτων, ε, των συνδικάτων κτλ. Σε ό,τι αφορά το επιπρόσθετο πρωτόκολλο, στο οποίο αναφερθήκατε. Αυτό είναι ένα πολύ σοβαρό θέμα. Ε, θα σας παραπέμψω στο αρχικό κείμενο και θα σας παραθέσω ένα απόσπασμα. Μετά από σοβαρές ε, συζητήσεις με τους συναδέλφους χθε, χθες, ε, καταλήξαμε στο εξής, ότι η Τουρκία πρέπει να εξασφαλίσει ότι εφαρμόζει το εθνικό το, προς το πρωτόκολλο της Συμφωνίας Σύνδεσης και κάνει πρόοδο στην προσπάθεια εξομάλυσης των σχέσεων με την Κύπρο. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα συνεχίσει την ανασκόπηση και εξέταση της προόδου με βάση τα συμπεράσματα του Συμβουλίου της 11ης ε, Δεκεμβρίου του 2006. Αν θεωρείτε ότι αυτά είναι κινέζικα, αυτή η δήλωση του Δεκεμβρίου του 2006 αναφέρεται ουσιαστικά στον, στην εξομάλυνση των σχέσεων ε, με την Κύπρο στα πλαίσια της ενταξιακής πορείας της Τουρκίας. Ο κύριος Τάλερ αναφέρθηκε στις δηλώσεις Γκρουέσκη και Παπανδρέου. Πραγματικά έχουμε μια μοναδική ευκαιρία. Και πιστεύω ότι σε αυτό το κρίσιμο θέμα τελικά θα κάνουμε πρόοδο. Η Κομισιόν δεν σκοπεύει να κάνει καμία προσπάθεια διαμεσολάβησης για αυτό το θέμα της ονομασίας ε, στα Σκόπια. Το κάνει ο ΙΕ και ο διαμεσολαβητής του ΙΕ, ο κύριος Νίμιτς. Ο κύριος Κάτσιν αναφέρθηκε στο κοσυφοπέθιο και στις θεωρήσεις. Σας ευχαριστώ για την υποστήριξή σας για το θέμα των θεωρήσεων. Απάντησα ήδη για το θέμα της Βοσνίας Ερσεγοβίνη. Έχετε δίκιο ότι πρέπει ότι χρειαζόμαστε αισιοδοξία στην Νοτιοανατολική Ευρώπη ε, και γενικά στο τομέα της διεύρυνσης. Ένας ε, επίτροπος διεύρυνσης πρέπει να είναι επαγγελματία αισιόδοξο. Κυρία Λούνατσεκ, αναφέρθηκε στο κοσφοπέδιο. Νομίζω ότι της έχω απαντήσει. Για το θέμα των Ρώμα. Είναι ένα πολύ σοβαρό θέμα. Καταλαβαίνω τις ανησυχίες σας. Αλλά καταρχάς αυτό είναι θέμα των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του αρμόδιου επιτρόπου για την ασφάλεια, δικαιοσύνη και ελευθερία. Δεν είμαι σε θέση να σχολιάσω αυτό το θέμα, ε, γιατί το χαρτοφυλάκιό μου επιβάλλει αυτόν τον περιορισμό. Ο κύριο Στάνοκ αναφέρθηκε στο Μαυροβούνιο. Συμφωνώ με την αξιολόγησή του. Το Μαυροβούνιο όντω είναι μια επιτυχημένη ιστορία στα Δυτικά Βαλκάνια. Έχει προβλήματα βέβαια σε ό,τι αφορά τη διαφθορά, το έγκλημα και την, τα διοικητικά της προβλήματα που είναι πολλά. Παρ' όλα αυτά η χώρα σημειώνει πρόοδο και ακριβώς γι' αυτό και ακριβώς γι' αυτό προχωρεί στον ευρωπαϊκό της δρόμο, στην ευρωπαϊκή της πορεία. Ευχαριστώ τον Επίτροπο. Πάμε τώρα στο δεύτερο γύρο ερωτήσεων. Με τον κύριο Κασουλίδη. 1,5 λεπτό. Ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε. Κύριε Επίτροπε, κάθε χρόνο η Επιτροπή ως έκθεση αναφέρει τα ίδια. Σχεδόν τα ίδια. Δεν έγινε η παρέκταση του πρωτοκόλλου της Αγγέλης Ευρωπαϊκής της Τουρκίας, δεν έχει ομαλοποιήσει σχέση με την Δημοκρατία της Κύπρου και κάθε χρόνο ε, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, παροτρύνει την ε, Τουρκία να, κάνει, να το κάνει αυτό και δεν το κάνει η Τουρκία. Και τι θα γίνει, business as usual δεν τρέχει τίποτα. Τι έγινε, ποιο επιβάλλει, ποιο ορίζει του όρου και τι προποθέσει να διαπραγματεύσουν η Τουρκία ή η Ευρωπαϊκή Ένωση. Ευχαριστώ κύριε Κασουλίδη. 1,5 λεπτό. Thanks very much. Thank you for all the cooperation you have and do give to this committee. Σας ευχαριστούμε για την ε, συνεργασία σας. Και ξέρετε για ε, τη δουλειά σας τις αμέσως επόμενες εβδομάδες σας εύχονται καλή επιτυχία όχι μόνο στους Δημοκράτες, όλοι μας, όλοι μας. Καλύφθηκα από αυτό που άκουσα για την Τουρκία ε, για την Αρμενία είναι πάρα πολύ καλά μας τα είπατε. Όντως έχετε δίκιο όσον αφορά τη, τις συμμεταρρυθμίση στη δικαιοσύνη ε, και την συνταγματική μεταρρύθμιση. Σωστά επίσης τα είπατε όσον αφορά τις μηνύσεις που πλήσουν την ελευθερία της έκφρασης στην Τουρκία. Θα τα δούμε αυτά από κοντά σε λίγο που θα πάμε εκεί. Ξέρετε, οι Τούρκοι αυτό και με βρίσκουν και μου λένε ότι είναι πάρα πολύ σημαντική η υπόθεση η προσχώρησή τους. Για πέστε μου. Τώρα για το θέμα του πρωτοκόλου της Τουρκίας. Τι θα κάνετε όσον αφορά το Συμβούλιο. Ποιο είναι το πρόβλημα. Δεν είναι το πρόβλημα αυτός από τα κόμματα και τις κυβερνήσεις. Πρόβλημα δεν είναι εκεί και η κοινή γνώμη. Ο κ. Μπαϊκάλ σήμερα ε, είχε συνομιλήσει και επαφές μαζί σας και ε, υπήρξαν και κάποιες θετικές δηλώσεις σχετικά. Ευχαριστώ. Ο κύριος Λαντστορφ. Ενάμιση λεπτό. Σας ευχαριστώ <clears throat> κύριε Πρόεδρε. Πρώτα θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Επίτροπο για τα καθαρά λόγια που είπε για την ελευθερία του τύπου και αυτό για μας τους φιλελευθέρους είναι πράγματα απαραίτητα. Α, έχω μια άλλη ερώτηση τώρα και που ξεφεύγει λίγο από την έκθεση Ακούσαμε ε, για σχέδιο ΡΕΝ 1 και σχέδιο ΡΕΝ 2 μεταξύ Κροατίας και Σλοβενίας, την προσπάθεια συμφιλίωσης δηλαδή, και φαίνεται πως υπάρχει κάποια πρόοδος τώρα, κάτι που με ικανοποιεί. Ποια διδάγματα βγάζετε εσείς για το μέλλον από την προσπάθεια αυτή, από τη συνεργασία σας με τις χώρες των Δυτικών Βαλκανίων σε ό,τι αφορά τη μελλοντική ε, στρατηγική και βέβαια τις σχέσεις και με τη Ρωσία. Εν τέλει ένα σύντομο σχόλιο είπατε ότι προτίθεται να ανοίξετε τις διαπραγματεύσεις με την Μακεδονία. Μην αναμένετε, αυτό θα ήθελα να σας πω, μην αναμένετε μεγάλο ενθουσιασμό από τις χώρες μέλη και ιδίω από τη δική μου χώρα για το θέμα αυτό. Είναι θέματα σημαντικά αυτά της διεύρυνσης και χρειάζονται ακόμα πάρα πολύ συζήτηση. Ευχαριστώ. Η πρόεδρος της αντιπροσωπείας με την Τουρκία, η κυρία Φλότχα, έχει το λόγο. Ευχαριστώ, πρόεδρε. Όπως και η κυρία Ρόιτον, ε, προτιμώ ε, τα προφορικά λόγια παρά τα γραπτά. Α, τα όσα ακούστηκαν μου προξενούν ανατρίχιασμα. Γιατί υπάρχουν κάποιε μεταρρυθμίσεις που δεν έχουν ε, τελεσφορήσει και θα πρέπει να τονίσουμε ότι πρέπει να συνεχιστούν. Ε, από την άλλη βέβαια έγιναν κάποιε σημαντικέ πολιτικέ πρωτοβουλίε, ε, πολύ ενθαρρυντικές. Νομίζω ε, ότι πρέπει να το υποστηρίξουμε αυτό. Ίσως όχι να δείξουμε υπερβάλλοντα ζήλο, αλλά τουλάχιστον να αναγνωρίσει η Ευρωπαϊκή Ένωση αυτό το καθεστώ. Δηλαδή η υπογραφή της συμφωνίας του πρωτοκολου αρμενια Τουρκία. Ε, μια δύσκολη ιστορία και για τις δύο πλευρές. Δεν έχει τελειώσει αυτή η ιστορία. Πρέπει να την υποστηρίξουμε. Σκέφτομαι επίσης ε, την ε, διαδικασία εκδημοκρατισμού για να αντιμετωπιστεί ένα βασικό θέμα, το κουρδικό θέμα. Είναι ένα κομβικό σημείο αυτό. Νομίζω ότι πρέπει να δείξουμε την υποστήριξή μας και σε αυτή την πρωτοβουλία σας ε, ρωτώ να μου πείτε, ε, υπάρχουν κάποιες πρωτοβουλίες που θα μπορούσαμε να προωθήσουμε εμείς στην Ευρωπαϊκή Ένωση για να βοηθήσουμε αυτή τη διαδικασία που, όπως είπε ο κύριος Όουιτ, είναι πάρα πολύ σημαντική ε, σημαντική διαδικασία για όλους τους πολίτες της Τουρκίας, για το δημοκρατικό τους μέλλον. Ευχαριστώ την κυρία Φλότχα και τώρα το λόγο έχει για 1,5 λεπτό πάντα ο κύριος Χατζηγεωργίου. Να ευχαριστήσω και εγώ τον κύριο Ρεν για τον πολύ κόπο που έκαμε για αυτή τη δουλειά. Είπατε ότι δεν είναι κινέζικα η απόφαση του Συμβουλίου του 6 για την Τουρκία. Διερωτούμε να παίξω κι εγώ λίγο το ίδιο λογοπαίγνιο κύριε Ρεν εάν μήπω είναι κινέζικα για την Τουρκία και θα σας πω μια δήλωση χθεσινή του κυρίου Μπαγής ο οποίος είπε ότι όσοι αναμένουν, έχοντας διαβάσει την έκθεση σας έτσι, όσοι αναμένουν από την Τουρκία να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της, θα πρέπει πρώτα να εκπληρώσουν τις δικές τους. Νομίζω ότι με κάποιο τρόπο αυτή η δήλωση, ή μάλλον ξεκάθαρα, στέλνει τις αποφάσεις που καταγράφονται στην έκθεσή σας στον κάλαθο των αχρήστων. Το 2006 η Επιτροπή πρότεινε κάποια μέτρα, κάποιες κυρώσεις που οδήγησαν στο πάγωμα 8 κεφαλαίων προτίθεται η Επιτροπή να προτείνει κάποιες κυρώσεις για το γεγονό ότι η Τουρκία δεν υλοποιεί το πρωτόκολλο. Θέλω επίσης να θυμίσω την δίκη που έγινε στην Τουρκία ενάντια στο κυβερνών κόμμα της Τουρκίας που καταδίκασε το δικαστήριο το κυβερνών κόμμα παρακαλώ και του απέκοψε την χρηματοδότηση και θέλω να δω πόσο συνάδει αυτό με ένα κράτος δικαίου στο οποίο αναφερόμαστε προηγουμένως. Και κλείνω, θέλω να ξέρω αν παρακολουθεί η Επιτροπή την δίκη για την ανακάλυψη των δολοφόνων του Χραν Τικ. Ευχαριστώ αγαπητέ συναδέλφε και τώρα το λόγο έχει ο κύριος Μπέλντερ για 1,5 λεπτό. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ως Πρόεδρος της Επιτροπής της ε, Αντιπροσωπείας για τις σχέσεις με το Ισραήλ μας ενδιαφέρει, με ενδιαφέρει πολύ η σχέση μεταξύ Ισραήλ και Τουρκίας. Ρωτώ λοιπόν τον Επίτροπο αν μπορεί να μας πει λίγο περισσότερα για την σελίδα 28 της εκθέσεώς του όπου αναφέρεται στις αντιδράσεις της Τουρκίας απέναντι στην κρίση στη Γάζα. Είναι σύντομη η παράγραφος αυτή, δεν φαίνεται ωστόσο να αναφέρεται στις ε, σοβαρές υπερβολές που έγιναν και ότι ε, ευθύνη γι' αυτό φέρει ο ίδιος ο κύριος Ερντογάν. Και με ενδιαφέρει ακόμα και τα φαινόμενα, με ενδιαφέρουν επίσης τα φαινόμενα αντισημιτισμού που σημειώνονται σε μια χώρα της διεύρυνσης η Τουρκία θέλει να παίξει ρόλο ως διαμεσολαβητής σε θέματα της Μέσης Ανατολής, αλλά η στάση της αυτή δεν βοηθεί. Τέλος, η διάκριση σε βάρος χριστιανών εθελοντών και σχετικών οργανώσεων στην Τουρκία. Ελπίζω θα μας δώσετε κάποιες απαντήσεις. Ε, θα κάνω μια εξαίρεση για τους δύο συντονιστές των Σοσιαλιστών και του ΕΛΚΑ που μου ζήτησαν να μιλήσουν μετά. Ενώ είχα κλείσει τον κατάλογο, αλλά δεν μπορώ να τους αρνηθώ. Θα τους δώσω το λόγο λοιπόν, αλλά για 1,5 λεπτό παρακαλώ. Έχω ορισμένες ερωτήσεις. Ο κύριος Επίτροπος είπε ότι σε σχέση με την Άγκυρα Δύο ισχύουν οι αποφάσεις Συμβουλίου και Επιτροπής του 2005. Αυτό σημαίνει ότι τώρα τέλη του 2009 λύγει μια προθεσμία μέχρι τα Χριστούγεννα. Από εκεί και μετά, όταν θα τελειώσει η προθεσμία αυτή, νομίζω ότι είναι ενδιαφέρον το ερώτημα. Τι θα γίνει μετά. Ευχαριστώ κύριε Μπροκ. Ο κύριος Βιγγένιν. Ευχαριστώ κύριε Αλμπερτίνη. Κύριε Ρέιν. Εκτιμώ την εισαγωγική σας παρέμβαση, γιατί υπάρχει ένα μάθημα το οποίο μπορούμε να μάθουμε από τις δραστηριότητε σας από την εντολή που έχετε και την πολιτική διεύρυνση. Ότι επιτυγχάνει μόνο όταν υπάρχει συνένεση ε, για τα θέματα στις υποψήφιες χώρες και όταν η πολιτική διεύρυνση δεν, γίνεται, δεν πέφτει θύμα ε, εσωτερικών έτσι, διαφωνιών και εσωτερικής πολιτικής ε, και εδώ και στα κράτη-μέλη. Μετά τη συνθήκη της Λισαβόνας και μετά την επικύρωσή της, ε, ελπίζω ότι θα έρθουν καλύτερες μέρες για την πολιτική διεύρυνση. Ελπίζω ότι θα έχουμε την θεσμική ευελιξία να συνεχίσουμε τις εργασίες μας και θα έχουμε τη δυνατότητα να δώσουμε ελπίδα στις υποψήφιες χώρες. Ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα είναι σε θέση πραγματικά να τις υποδεχθεί και όχι μόνο να συνομιλεί μαζί τους. Επίσης εκτιμούμε και το θέμα αυτό για την απελευθέρωση της υποχρέωσης θεωρήσεων, γιατί είναι ένα σοβαρό κίνητρο για τους κατοίκους περιοχής να συνεχίσουν προσπαθίες τους. Μια γενική ερώτηση. Ποια είναι η εκτίμησή σας. Μπορούμε να πούμε ότι τώρα οι υποψήφιες χώρες είναι πιο κοντά στην εκπλήρωση των προϋποθέσεων σε σχέση με την κατάσταση που επικρατούσε πριν από ένα <coughs> χρόνο. Και ποιε είναι οι προβλέψει σα για τα επόμενα πέντε χρόνια, πολύ σύντομα. Και ένα ειδικό ερώτημα για την Τουρκία. Ποια είναι η γνώμη σα για τα μεικτά μηνύματα που τη στέλνουμε της Τουρκίας. Και μία παρατήρηση. Εκτιμούμε τη συμφωνία που υπογράφηκε μεταξύ Τουρκίας και Αρμενίας. Πώς εκτιμάτε όμως ότι υπογράφτηκε σε μια χώρα που δεν είναι ε, μέλος Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και η, η, το, η στάρ αυτή που πρωταγωνίστησε στην όλη διαδικασία ήταν η Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών. Διακόπτει όμως ο Πρόεδρος. Πρώτα, συγχαρητήρια κύριε Ρέν για την ανεκτική, δημιουργική και ειρηνική αντιμετώπιση των προβλημάτων. Σε εποχή όπου το πρόβλημα του εθνικισμού προκαλεί ναι, ο εθνικισμός προκαλεί ακόμα σημαντικά προβλήματα. Ελπίζω σε μικρότερο βαθμό σιγά σιγά στην περιοχή αυτή του κόσμου και είναι βέβαια καθήκον της Ευρωπαϊκής Ένωσης να αντιμετωπίσει και το πρόβλημα αυτό. Συγχαρητήρια λοιπόν για το τμήμα αυτό της έκθεσής σας που αναφέρεται στο άνοιγμα των διαπραγματεύσεων με τη Μακεδονία. Θα χρειαστεί πολύ καλή θέληση και συμπάθεια προς την χώρα αυτή για να μπορέσει να ξεπεραστεί το πρόβλημα της ονομασίας. εκφράζω την ικανοποίησή μας στο όνομα της ομάδας των φιλελεύθερων και για τις διαπραγματεύσεις με την Κροατία που μπαίνουν σε καλή φάση. Μένουν τρία ανοιχτά προβλήματα τα οποία πρέπει να αντιμετωπιστούν. Η επιστροφή του σερβικού πληθυσμού, το, η εγκληματικότητα και βέβαια τέλος τα ανοιχτά προβλήματα στα σύνορα με άλλες χώρες. Για το Μαυροβούνιο το ανοιχτό ερώτημα είναι βέβαια ακόμη το οργανωμένο έγκλημα και η, άσκηση, και, συγγνώμη, και η πίεση που ασκείται στα μέσα ενημέρωσης. Ευχαριστώ. Κλείνουμε το δεύτερο γύρο ερωτήσεων με την κυρία Κοπά για, τα, για 1,5 λεπτό. Ε, thank you, President, ε, Mr. Commissioner. you very σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, σας ευχαριστώ κύριε Επίτροπε. Έχω λίγα σύντομα σχόλια. Οι πρόσφατες εκλογές στην Ελλάδα και η επιστροφή του Γεωργίου Πανδρέου ως Πρωθυπουργού και Υπουργού Εξωτερικών δίνουν ε, σημαντικές ελπίδες για την αναζαγόνηση της ε, ατζέντα Θεσσαλονίκη και ίσως μάλιστα να προχωρήσει και ένα βήμα παραπέρα. Η νέα κυβέρνηση ασφαλώς ενδιαφέρεται να προωθήσει τις διαπραγματεύσεις αλλά όπως γνωρίζετε για να χορέψουν ταγκό χρειάζονται δύο. Άρα χρειάζεται μια αμοιβαία αποδοχή συμφωνία. Ελπίζουμε ότι η Κομισιόν θα βοηθήσει. Διότι η ε, επίλυση του προβλήματος αυτού είναι απόλυτη προϋπόθεση για την Ελλάδα για να μπορέσει να προχωρήσει η υπόθεση. Τώρα, για την Τουρκία. Επανήλθε στην Τράπεζα των Διαπραγματεύσεων. Αλλά η απογοήτευσή μου οφείλεται στο γεγονός ότι δεν γίνεται αναφορά στο γεγονός ότι η χώρα αυτή δεν τηρεί τις διμερείς συμφωνίες που συνυπέγραψε με την Ελλάδα το 2002, κάτι το οποίο προκαλεί πολλά προβλήματα, όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ποια είναι η θέση σας λοιπόν σχετικά με την υποχρέωση της Τουρκίας να τηρήσει την συμφωνία αυτή. Και τώρα ε, δύο τελευταία λόγια για τη Σερβία. Είναι θετικό που η μονομερής εφαρμογή της ε, προσωρινής συμφωνίας περιλαμβάνεται μέσα στην συμφωνία, στην ε, έκθεση μάλλον. Μέχρι τώρα όμως το Συμβούλιο δεν έχει συμφωνήσει να κάνει σχετική αναφορά. Μπορούμε να περιμένουμε ε, τέτοια αναφορά στα συμπεράσματα του Συμβουλίου του Δεκεμβρίου. Ευχαριστώ. Κλείνουμε έτσι το δεύτερο γύρο παρεμβάσεων, ερωτήσεων και τώρα έχει το λόγο ο Επίτροπος για να απαντήσει. <clears throat> Σας ευχαριστώ για τις ενδιαφέρουσες ερωτήσεις σας. Θα προσπαθήσω να τις ομαδοποιήσω ώστε να δώσω πιο ξεκάθαρες απαντήσεις. Πρώτα, για το πρωτόκολλο της Αγκύρας που έθεσε ο κύριος, ο κύριος Κασουλίδης, ο κύριος Χατζηγεωργίου, ο κύριος Μπροκ, αλλά και ο κύριος Χόιτ έφυξε το θέμα και ορισμένοι άλλοι. Ασφαλώς το θέμα είναι από αυτά που έχουν προτεραιότητα. Σύμφωνα με τα συμπεράσματα του Συμβουλίου του Δεκεμβρίου του 2006 υπενθυμίσατε άλλωστε ότι έχουμε αναστείλει οκτώ κεφάλαια στις διαπραγματεύσεις με την Τουρκία. Από ένα σύνολο 35. Οκτώ σημαντικά κεφάλαια. Για παράδειγμα, εξωτερικές οικονομικές σχέσεις, γεωργία, μεταφορές και άλλα. Λόγω της μη συμμόρφωσης της Τουρκίας με το πρωτόκολλο της Αγγίρας Εκτός αυτού, μία χώρα μέλος μπλοκάρει στην ουσία πέντε κεφάλαια. Μια άλλη χώρα μπλοκάρει στην ουσία πολλά άλλα κεφάλαια. Και αυτά τα πράττουν για διμερείς λόγους ή πάντως όχι για λόγους που να έχουν συμφωνηθεί με τους άλλους. Έχουμε βέβαια και τα benchmarks για να ανοίξουμε και άλλα κεφάλαια. Αν τα πράγματα μείνουν όσοι έχουν, θα μας τελειώσουν τα κεφάλαια πολύ σύντομα ο θεσμικός μας ρόλος ως Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι να κάνουμε μια αντικειμενική αξιολόγηση. Το πράξαμε αυτό, είπαμε και επικρίναμε την Τουρκία για την μη πλήρη εφαρμογή του πρωτοκόλλου της Το Συμβούλιο τώρα θα πρέπει να συναγάγει τα συμπεράσματά του και να λάβει τις σχετικές αποφάσεις. Αυτά θα τα συζητήσει το Συμβούλιο θα τα συζητήσει το Συμβούλιο τον Δεκέμβριο και για το ειδικότερο αυτό θέμα. Η διατύπωση των συμπερασμάτων του Δεκεμβρίου 2006 είναι ακόμα ανλοπή στη μνήμη μου γιατί τα είχα γράψει εγώ ίδιος και έχουν ως εξή. Απ' έξω τα ξέρω. Στα επόμενα χρόνια η Κομισιόν και το Συμβουλίο θα εξετάσουν την πρόοδο της Τουρκίας σε σχέση με την εφαρμογή του πρωτοκόλου της Αγκύρας. Στα επόμενα χρόνια και ιδίως το 2007, 2008 και μέχρι το 2009 βάλαμε και αυτά τα χρόνια γιατί ορισμένες χώρες μέλη είχαν εκλογές τα χρόνια αυτά. Δεν σημαίνουν όμως ότι πρόκειται για προθεσμία ότι δηλαδή λύγει κάποια προθεσμία τον Δεκέμβρη του 2009. Αναφέρθηκαν τέτοια αυτά περισσότερο ενδεικτικά, 07, 08 και 09. Αυτή είναι η κατάσταση. Πάντως πρέπει να τονιστεί και πάλι η σημασία της υποχρέωσης αυτής της Τουρκίας να εφαρμόσει πιστά το πρωτόκολλο της Αγγίρας και θα τα περιλάβουμε στα συμπεράσματά μας αυτά και είναι και σημαντικό μέτρο αποκατάστασης εμπιστοσύνης να υποστηρίξουμε δηλαδή τις διαπραγματεύσεις ώστε αυτές να μπορέσουν να απολύξουν εν τέλει σε μια επανένωση της νήσου Κύπρου και να μπορέσει η Κύπρος να γίνει επιτέλους μια χώρα μέλος η οποία να μπορεί να ε, λειτουργήσει φυσιολογικά ενωμένη. Όταν, μπαίνω, όταν φτάνω στην Λευκοσία έχω την εντύπωση ότι μπαίνω σε μια χρονομηχανή και επιστρέφω στις εποχές του Checkpoint Charlie στην ε, Γερμανία γιατί υπάρχουν τόσες ε, φυλασσόμενες διαβάσεις για τα σύνορα και τα ανάμεσα στην πράσινη γραμμή δηλαδή και ούτε καθεξής. Τώρα, για το κουρδικό. Επίσης ένα σημείο εστίασης και σημαντικό θέμα εσωτερικής πολιτικής στην Τουρκία. Θα αντιληφθήκατε ότι οι απόψεις μας είναι γνωστές στην Τουρκία. Εμείς ζητούμε πολιτιστικά και γλωσσικά δικαιώματα υπέρ όλων των πολιτών τουρκικής καταγωγής και των ε, κουρδικής προέλευσης. τους τελευταίους μήνες πήγαν ορισμένα πράγματα καλύτερα στην Τουρκία και είχαμε λόγους να εκφράσουμε κάποια ικανοποίηση. Φέτος άνοιξε ένας σταθμός τηλεόρασης με 24 ώρες το 24ωρο εκπομπές σε κουρδική γλώσσα και εθνικό κανάλι αυτό. Αναμένουμε και άλλες πρόοδους τέτοιες βασισμένες σε μια ευρεία διαβούλευση που έχουν ως στόχο να αυξήσουν τα πολιτιστικά δικαιώματα σε θέματα όπως η εκπαίδευση, η πρόσβαση άλλωστε σε δημόσιες υπηρεσίες κλπ. Στην έκθεσή μας λέμε ότι η Τουρκία πρέπει να διασφαλίσει πολιτιστική διαφοροποίηση και προστασία μειονοτήτων και όλων των πολιτών ανεξαρτήτως καταγωγής. Θεμελιώδη ανθρώπινα δικαιώματα είναι αυτά. Ο Γιος Χόουιτ αναφέρθηκε στις σχέσεις μεταξύ Τουρκίας και Αρμενίας. Απάντησα ήδη εν μέρη σε σχέση με την εξομάλυνση των σχέσεων αυτών και νομίζω ότι είναι πάντως ενδιαφέρον να αναφερθώ και στην εκστρατεία Τούρκων διανομένων για να αλλάξει η στάση απέναντι στη σφαγή των Αρμενίων του 1915. Θέμα ιδιαίτερα οδυνηρό, βέβαια, για όλους. Το πρώτο, το πρώτο μας μήνυμα είναι σε αυτές τις περιπτώσεις να ζητήσουμε, σε την περίπτωση δηλαδή να ζητήσουμε ειλικρινή διάλογο. Έχουμε βαθύτατο σεβασμό για την ιστορία και για την μνήμη των ανθρώπων που έχασαν τη ζωή τους εκείνα τα χρόνια του 1915. Είναι πάντως κάτι το οποίο πρέπει να εξεταστεί μέσα σε σοβαρό επιστημονικό πλαίσιο από τους ιστορικούς με πλήρη ελευθερία. Και γι' αυτό είναι σημαντικό να φτάσει έχει φτάσει μάλλον η ελευθερία έκφρασης άποψης στην Τουρκία σε ένα επίπεδο όπου οι Τούρκοι διανόμενοι μπορούν να ε, εκφράσουν άποψη πλέον και για το θέμα αυτό. Θα πρέπει να φροντίσουμε και αυτήν την ε, επούλωση των πληγών του παρελθόντος που γίνεται σε εθνικό επίπεδο και βέβαια και απέναντι στην Αρμενία. Η ερώτηση του κ. Λάμπστορφ ρώτησε ποια διδάγματα αντλούμε για το μέλλον από την ε, σύγκρουση μεταξύ των χώρων Κροατίας και Σλοβενίας για συνοριακές διαφορές. Αναμίχθηκα πολύ έντονα στην εργασία αυτή μεταξύ Ζάγκρεπ και Λουμπλιάνας σε μια προσπάθεια που αρχικά είχε λήξει τον Ιούνιο με την τελευταία μου πρόταση για μια συμφωνία διατησίας είχε υποβληθεί στις δύο χώρες. Είχαν μείνει κάποιες λεπτομέρειες, δύο λέξεις ήταν τρεις, ενώ είχαμε ξεκινήσει από μεγάλη απόσταση. Η Σλοβενία ζητούσε πολιτική συμφιλίωση είχε ακουστεί και το όνομα του Μάτι Αχτισάρη ως ενδεχόμενο μεσολαβητού ενώ η Κροατία ζητούσε να υπαχθεί το θέμα στο Διεθνές Δικαστήριο. Εμείς προτείναμε Διεθνές Διεθνικό Δικαστήριο που είναι διεθνές όργανο αλλά έχει και διαμεσολαβητικό ρόλο μετά από τη δική μου διαμεσολάβηση. Οι δύο πρωθυπουργοί μπόρεσαν να συνεργαστούν και να αποκαταστήσουν, αμοιβαία εμπιστοσύνη και με κάποια τεχνική υποστήριξη της Κομισιόν μπόρεσαν να προχωρήσουν και να ξεμπλοκάρουν έτσι οι διαπραγματεύσεις Ένταξη τη Κροατία προ 15 μέρου. Ένα δίδαγμα για το μέλλον πάντως ήταν ότι δεν είναι εύκολο για την Κομισιόν να μεσολαβήσει ανάμεσα σε μια ήδη χώρα μέλος και σε μια χώρα η οποία βρίσκεται υπό ένταξη. Γιατί υπάρχει πάντοτε η υποψία ότι η ε, Κομισιόν θα ταχθεί περισσότερο υπέρ της χώρας μέλους. Βέβαια υπάρχει κοινωνική προτίμηση και ε, είμαστε υποχρεωμένοι να φροντίσουμε ε, τα συμφέροντα των χωρών μελών μας. Άρα η αφετηρία μας δεν ήταν πάρα πολύ καρποφόρα, αλλά τώρα εν πάση περιπτώσει έχουμε μια συμφωνία και ελπίζω ότι από εδώ και μπρος οι σχέσεις των δύο χωρών θα είναι πιο θετικές. Σε ό,τι αφορά ακόμη τα διδάγματα για την εξωτερική πολιτική, νομίζω ότι στην ουσία υπάρχουν τρία διδάγματα. Πρώτα, η θεμελίωση της κοινή εξωτερικής πολιτικής θα πρέπει να είναι τέτοια που να προβάλλει την σταθερότητα στην γειτονιά μας που είναι οι χώρες των Βαλκανίων η Μεσόγειος, η Νοτιοανατολική Ευρώπη, ώστε να είμαστε αξιόπιστοι ως παγκόσμιος παίκτη. Αν δεν μπορούμε να συμβάλλουμε στην σταθερότητα στην γειτονιά μας, στην αυλή μας, πώς να αναμείνουμε να είμαστε αξιόπιστοι αλλού. Γι' αυτό η συνέχεια και η αξιοπιστία της ε, ε, πολιτικής διεύρυνσης είναι πολύ σημαντικές. Τώρα, η, τα ισχυρά σημεία της ενιαίας αγοράς, όπως η περιβαλλοντική νομοθεσία, προστασία του καταναλωτού, πρέπει να είμαστε περισσότερο ικανοί να μεταφέρουμε αυτά τα εσωτερικά ισχυρά σημεία μας και προς τις εξωτερικές σχέσεις. Να τα εμφανίσουμε ως ευρωπαϊκές αξίες να τα βάλουμε στην βάση της προσπάθειας υποστήριξης και υπεράσπισης των ευρωπαϊκών συμφερόντων μέσω των πολιτικών μας. Παράδειγμα, ενέργεια. Που θα είναι από τα πιο σημαντικά θέματα και για την επόμενη Επιτροπή και για το Κοινοβούλιο. Στον τομέα της ενεργειακής πολιτικής, όπου ο Επίτροπος Πίμπαλξ έχει ε, επιτελέσει σημαντικό έργο, και χρειάζεται βέβαια και η ενιαία αγορά εκεί γιατί αυτή είναι η βάση της ε, σταθερότητας γιατί μπορείτε να φτιάξετε αγωγούς από εδώ και από εκεί αλλά το θεμέλιο δεν μπορεί παρά να είναι η ενιαία αγορά και η διασυνδέση μεταξύ των χωρών. Και τέλος πρέπει να εκμεταλλευτούμε κάθε ευκαιρία που δίνει η συνθήκη της Λισαβόνας να χρησιμοποιήσουμε τους νέους μηχανισμούς που προσφέρει για, την, για να δώσει κατευθύνσεις στην εξωτερική πολιτική. Μελετώ προσεκτικά την έκθεση του Έλμαρ Μπροκ και χαίρομαι που το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο συζητεί ενεργά το θέμα και λαμβάνει θέση. Βρισκόμαστε στην ίδια λέμβο, αν μπορώ να το πω έτσι. Και πρέπει να συμβάλλουμε όλοι. γιατί και η συνθήκη της Λισαβόνας σας προσφέρει εσάς, σε εσά στην Επιτροπή Εξωτερικών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σημαντικότερο ρόλο και είμαι πεπισμένο ότι θα μπορέσετε να εκμεταλλευτείτε τις ευκαιρίες αυτές με σόφρονα τρόπο. Τώρα πάμε στο τελευταίο γύρο ερωτήσεων. Έχουμε ακόμα 10 ομιλητές. Δυστυχώς, θα πρέπει να σας περικόψω κι άλλο το χρόνο, σε ένα λεπτό. Ο κύριος Θεοχάρους, η κυρία Θεοχάρους, έχει το λόγο. Ευχαριστώ. Έχω δύο ερωτήσεις. Για την ε, Βοσνία είπατε ότι δεν μπορεί ένα προτεκτοράτο να μπει στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Να συμπεράνουμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν θα δεχθεί τους όρους της Τουρκίας για το αναχρονιστικό θεσμό των εγγυήσεων όσον αφορά την Κύπρο που θα μετατρέψουν ένα ανεξάρτητο κράτος σε προτεκτοράτο. Η δεύτερη ερώτηση. Είπατε ότι, μάλλον στην έκθεση αναφέρεται ότι η Τουρκία στηρίζει τις συνομιλίες και ότι δεν υπάρχει καταληκτικό όριο το 2009. Σας λέγω ότι η Τουρκία στηρίζεται συνομιλίες μόνο όταν διεξάγονται κάτω από τους όρους που θέλει η ίδια και προς την κατεύθυνση που θέλει η ίδια, δηλαδή της διχοτόμησης και των δύο κρατών να υποθέσουμε ότι ενώ αναγνωρίζεται πως δεν έχει προχωρήσει σε εξομάλυση των σχέσεων με την Κύπρο, δεν προτείνεται κυρώσει για να μην κατηγορηθεί η Κομισιόν ότι τάσεται υπέρ της Κύπρου και σε βάρος της Τουρκίας, όπως αναφέρατε τώρα στην τελευταία αποστροφή της δηλωσή ε, δήλωσής σας. Ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα να πω πολύ περισσότερα, αλλά... Ε, και τώρα, ο κύριος Κυρίλοφ, ένα λεπτό. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Επίτροπε. Πρέπει να σας συγχαρούμε για την εκθεσή σας. Αυτό που είναι σημαντικό είναι ότι κρατάμε ανοιχτή την προοπτική για όλες τις χώρες των Δυτικών Βαλκανίων. Σε ό,τι αφορά την Μακεδονία, είναι καλό που ξεκινήσατε την έναρξη. Θα δούμε πότε θα ξεκινήσει πραγματικά η ενταξιακή διαδικασία, αλλά όταν ξεκινήσει θα πρέπει να καταλάβει η Μακεδονία ότι θα υπάρξει παρακολούθηση του σύνεγγυ όταν ξεκινήσουν οι διαπραγματεύσει. Θα πρέπει να χαιρετήσουμε βέβαια το γεγονός ότι μπορούν τώρα οι Μακεδόνες να ταξιδεύουν ελεύθερα χωρίς θεωρήσεις ε, και θα μπορούν να ταξιδεύουν ελεύθερα και στην Ελλάδα και αλλού. Είναι πολύ σημαντικό η κυβέρνηση της Μακεδονίας να γνωρίζει ότι η οικοδόμηση καλής ε, γειτονίας και η οικοδόμηση ενός έθνους δεν έχει καμία σχέση με τις χειραγωγήσεις του, της ιστορίας του παρελθόντος, της ιστορίας και του παρελθόντος. Ε, όλα αυτά είναι τελείως διαφορετικά πράγματα. Ο κύριος Γκέρενς για ένα λεπτό. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Α μιλήσουμε για την αξιοπιστία τη ε, διαδικασία ε, διεύρυνση τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Για να είμαστε αξιόπιστοι, αυτή η διαδικασία θα πρέπει να έχει δύο μέρη ε, που σέβονται τι δεσμεύσει του. Οι χώρε που θέλουν να ενταχθούν στην Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να σεβαστούν τι δεσμεύσει του, θα πρέπει να υπάρχει η σύμφωνη γνώμη του Κοινοβουλίου και θα πρέπει και όλα τα κράτη-μέλη τη Ευρωπαϊκή Ένωση να συμφωνήσουν. Όμω μέχρι πρότινος η επικύρωση της ε, συνθήκης της ε, Λισαβόνας είχε δημιουργήσει ε, εχθρότητες στην ενταξιακή συγγνώμη, διαδικασία από πολλές χώρες. Τώρα που αλλάζουν τα πράγματα για την Λισαβόνα, μπορείτε να πείτε ότι όλες οι επιφυλάξεις των κρατών μελών έχουν αρθεί για την διεύρυνση. Ναι ή όχι. Ευχαριστώ το λόγο για ένα λεπτό η κυρία Κορνελίσε. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Πάρα πολύ ενθαρρυντικά αυτά, πάρα πολύ αξιέπαινα το ότι ε, έβαλε η Ελλάδα στην άκρη αυτέ τι εθνικέ συζητήσει, ώστε να βοηθήσει στην ε, ευρωπαϊκή πορεία της... Ε, Μακεδονία, τουλάχιστον στα πλαίσια Ευρωπαϊκή Επιτροπή, όμως τελικά το Συμβούλιο θα αποφασίζει αν, κατάλαβα καλά κύριε Ρεν, είπατε ότι εύχεστε να, αναλυθεί το, πρόβλημα πριν να ε, ληφθεί η απόφαση ή θα, και θα εξαρτηθεί τόσο πάντων από το, από το, το, αν θα επιληθεί το πρόβλημα, το τι θα αποφασίσετε εσείς. Ε, στη Βοσνία φυσικά τα πράγματα ε, βρίσκονται σε κατάσταση εμπλοκής και ε, έχουμε ποντάρει στις συνομιλίε που τώρα λαμβάνουν χώρα όμως δεν νομίζω ότι εκεί υπάρχει η κατάλληλη προπαρασκευή και έτσι δεν υπάρχει μια ιδιαίτερη συμβολή. Για πέστε μου. Ευχαριστούμε κύριε Κορνέλη, είναι Και τώρα. Έχετε το λόγο κύριε Μέντλε. Το προηγούμενο Σαββατοκύριακο πρόεδρε στην πατρίδα μου στις κάτω χώρες μια ομάδα Ρουμάνων παραλίγο να με ληστέψουν. Εσείς τι λέτε, μια που είσαστε υπεύθυνο κύριε Ρέν, κύριε Ρέν σε εσάς το λέω, για το ότι η Ρουμανία μπήκε στην Ευρωπαϊκή Ένωση και εμείς έχουμε γίνει θύματα εγκληματικών του ενεργειών. Τι, άρα, τι, πού το πάτε, ε? θέλετε κι άλλες διευρύνσεις. Και γιατί νομίζετε ότι η Τουρκία διατυπώνει όλα αυτά τα αιτήματα ενταξή. Είναι Ισλαμική χώρα. Από όλου μα εδώ είσαστε ο πιο αφελεί γιατί δεν μπορείτε να διαπιστώσετε ότι αυτή τη στιγμή το Ισλάμ είναι μια ιδεολογία. Και ε, είναι πάλι ένα, θέμα του, του πώ θα Λα πάρει τη θέση της πολιτικής στο μυαλό των προσώπων. Τώρα, για την ε, Κύπρο δεν ξέρω τι θα γίνει. Θα πάω στην ε, Άγκυρα κι εγώ και ε, θα ήθελα να έχω μια επιστολή μαζί μου δική σας που να λέει ότι μέχρι το τέλος της χρονιάς θα αποσυρθεί η, Κύπρος, η Τουρκία από την Κύπρο. Αυτό είναι το πάω στον Ερντογάν. Ευχαριστούμε, λέει ο Πρόεδρος. Και τώρα. Μαύρο Νικόλας. Σε πλήρη αντίθεση σε σχέση με την έκθεση προόδου της Τουρκίας και πολύ δε περισσότερο που φαίνεται να υποβαθμίζονται από τον κύριο Επίτροπο τα ιστορικά ραντεβού του 6, του 7, του 8 και σήμερα του 9 χωρίς να αφήνεται περαιτέρω περιθώριο για διερεύνηση των προθέσεων της Τουρκίας σε σχέση με το μεγάλο θέμα του κυπριακού προβλήματος. Θεωρώ ότι το κυπριακό πρόβλημα είναι ευρωπαϊκό πρόβλημα. Θεωρώ ότι ασχολούμαστε με τα ανθρώπινα δίκαια για τον τελευταίο πολίτη ανά το παγκόσμιο. Οφείλουμε να ασχοληθούμε πραγματικά με το κυπριακό πρόβλημα. Λαμβάνοντα υπόψη ότι σήμερα όχι μόνο δεν βοηθεί τις συνομιλίε, η Τουρκία αλλά μιλά για δύο κράτη, λαμβάνοντα υπόψη ότι σήμερα η Τουρκία συνεχίζει τον επικισμό των κατεχομένων και έχουμε 400.000 έπικους σε έναν πληθυσμό ενό εκατομμυρίου. Άρα με αυτά τα δεδομένα η έκθεση δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα. Δεν έχω καμία ερώτηση για τον κύριο Επίτροπο. Ευχαριστώ τον κύριο Μαυρονικόλα. Βαν Μπάλεν, ένα λεπτό. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Και εγώ είμαι από την Ολλανδία με τον προηγούμενο, όπως και ο προηγούμενος ομιλητής, αλλά ποτέ δεν έκλεψε κανένας Ρουμάνος. Θέλω να το πω από την αρχή. Μία ερώτηση προς τον κύριο Ρέιν. Ο κύριος Ρέιν είπε ότι είναι αισιόδοξο, ε, μια και είναι επίτροπος διεύρυνσης. Εγώ θα ήθελα να είμαι ρεαλιστής καλύτερα παρά αισιόδοξο. Η Τουρκία δεν θέλει να επικυρώσει και να εφαρμόσει το πρωτόκολλο της Άγκυρας. Ο Υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας έφτασε, ήρθε πρόσφατα στην Ολλανδία και έδωσε και μία συνέντευξη. Υπάρχει μάλιστα ε, και απόσπασμα της συνέντευξής του και είπε ότι δεν θα το εφαρμόσουμε γιατί το βόρειο τμήμα της Κύπρου δεν θα, πρέπει, να απομονωθεί περαιτέρω. Νομίζω ότι πρέπει να επικυρώσει και να εφαρμόσει το πρωτόκολλο. Τι θα κάνουμε εμεί για να αναγκάσουμε την Τουρκία να το κάνει. Θα ήθελα, Επίτροπε, να μου δώσετε μια ξεκάθαρη απάντηση. Θα παγώσουν διαπραγματεύσει ή υπάρχουν άλλε κυρώσει που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε. Κύριος Μούνιτς. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε και ευχαριστούμε κύριε Επίτροπε. Είναι πολύ σημαντικό να συνεχίσει η πρόοδο τη ε, διαπραγματεύσει τη ε, διεύρυνση και μου φαίνεται ότι είναι πάρα πολύ ικανοποιητική η κατάσταση ε, που διέπει τώρα την κατάσταση που είναι τόσο περίπλοκη στο κοσυφοπαίδιο. Θα πρέπει τα κεφάλαια να μείνουν ανοιχτά, σωστά, έχουμε άρετες τους περιορισμούς της θεωρήσει διαβατηρίων και τώρα έχουμε τα θέματα τα φορολογικά που ε, περνάνε από τις διαπραγματεύσεις και επίσης θα πρέπει ε, να προχωρήσουμε σύμφωνα με το 1244 το ψήφισμα του ΟΗΕ και με όλο το σεβασμό με τους συναδέλφους που είναι αναπληρωτές εδώ ε, είναι κακό διότι όταν τόσο πολλοί ζητούν το λόγο τελικά δεν μπορούν τα τακτικά μέλη να μιλήσουν όσο θέλουν. Αυτό προσπαθήσαμε να κάνουμε πάντως, να εξασφαλίσουμε. Ε, η κυρία Μπόσκουρτ, ένα λεπτό. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα ήθελα να θέσω ένα ερώτημα για τη Βοσνία. Ως ε, σκιώθηση γήτρια για τους σοσιαλιστές. Μιλήσατε για το αδιέξοδο που υπάρχει στη Βοσνία. Τι περιμένετε από τις συνταγματικές μεταρρυθμίσεις γιατί η διαδικασία λήψης των αποφάσεων ε, στη χώρα αυτή ε, συναντά δυσκολίε. Μήπως αυτά που λέμε εμείς εδώ πέρα είναι απλώς ευχολόγια. Μια άλλη ερώτηση. Ότι τα διμερεί θέματα δεν θα πρέπει να προκαλέσουν προσκόμματα στη διαδικασία διεύρυνσης, όπως ας πούμε στην ε, Κροατία. Στην περίπτωση της Τουρκίας όμως υπάρχουν τέτοια προβλήματα. Τα διμερεί θέματα δημιουργούν προσκόμματα στην ε, διαδικασία ένταξη. Μπορείτε να μου το εξηγήσετε αυτό, γιατί νομίζω ότι αντιφάσκεται λιγάκι εδώ πέρα. Ευχαριστώ την κυρία Μπόσκουρτ. Παντσέρη, ένα λεπτό. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Μία απλή ερώτηση, γενική φύσεω. Βλέπω τα στοιχεία πρόοδου, αλλά υπάρχουν και κάποια σημεία που εγείρουν αμφιβολίες. Νομίζω αν θέλουμε να επιλύσουμε το βαλκανικό θέμα, ε, πρέπει να το καταλάβουμε. Θα πρέπει να έχουμε μια συνολική εικόνα της περιοχής και όχι μια ε, εικόνα κατακαιρματισμένη. Ε, ενδεχομένως όμως αν αντιμετωπίσουμε συνολικά τις χώρες αυτές μπορεί να οδηγηθούμε σε καθυστέρηση της ενταξιακής διαδικασίας. Αν α, τις κοιτάξουμε κατακαιρματισμένα μπορεί κάποιες χώρες να μείνουν απ' έξω να χάσουν το τρένο. Ε, τι έχετε να μου πείτε για αυτή την, την άποψη. Ε, πώς βλέπετε το, τη σκέψη αυτή. Διμερής προσέγγιση ή συνολική. Ευχαριστώ. Φεζό. Ένα λεπτό. Ε, καλωσορίζω τα όσα μας είπε ο Επίτροπος για τα Δυτικά Βαλκάνια. Ως εισηγήτρια για την διαδικασία απελευθέρωσης από την υποχρέωση θεωρήσεων για τα Δυτικά Βαλκάνια, θα ήθελα να σας κάνω έκκληση να σεβαστείτε τις αυστηρές προϋποθέσεις και για την Βοσνία ε, Ερσεγοβίνη και για την Αλβανία. Δεν πρέπει να γίνουν ο... όμοιροι αυτές οι δύο χώρες ε, της όλης διαδικασίας. Πότε πιστεύετε να ταξιδέψουν οι άνθρωποι ελεύθερα, οι άνθρωποι αυτών των περιοχών, της Βοσνίας, εσεγοβίνης ε, του Κοσφοπεδίου κτλ. Και για την Κροατία ε, υπάρχουν διάφορα ανεπίλητα θέματα. Όπως παραδείγματο χάρη της τράπεζας της α, Λουμπλιάνας. Τι έχει γίνει με αυτό το θέμα. Εκτός καταλόγου, για ένα λεπτό, Κύριος Παπα-Νικολάου. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε. Ε, δεν είμαι μέλος αυτής της Επιτροπής, αντικαθιστώ όμως την κυρία Γιαννάκου και τον κύριο Κουμουτσάκο. Σε ό,τι αφορά την Τουρκία, αναφέρθηκαν οι δυσκολίες για την, για την ένταξη. Ε, παρά την περιγραφή των αδυναμιών όμως, δεν, υπάρχουν, δεν υπάρχει στην έκθεση πρόβλεψη κυρώσεων. Και ρωτώ για ποιο λόγο συμβαίνει αυτό και αν σκοπεύει η Επιτροπή να κάνει μια σχετική εισήγηση προ αυτή την κατεύθυνση στο Συμβούλιο. Και σε ό,τι αφορά τα Σκόπια, την γειτονική μα χώρα, τη οποία καλωσορίζουμε την πρόοδο και για την οποία υπενθυμίζω ότι η ονομασία τη, η επίσημη, η διεθνή ονομασία τη είναι Former Euro, ε, Yugoslavian Republic of Macedonia και όχι άλλε αναφορέ που έγιναν, ρωτώ σε σχέση με την διεύρυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συμπεριφορές εθνικιστικού χαρακτήρα σε μια Ευρώπη της πολιτισμικότητος είναι θεμητές. Ποια η άποψή σας γι' αυτό. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ κύριε Παπα-Νικολάου. Έχουμε λίγη ώρα ακόμα στη διάθεσή μας. Πριν έρθει εδώ η Επιτροπή, Υποεπιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, άκουσαμε πολλοί άριθμες ερωτήσεις. Ο λόγος στον Επίτροπο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ας ξεκινήσουμε με τα όσα είπε ο κύριος ε, Μαυρονικόλας, Φαν Μπάλεν, Θεοχάρος και Παπα-Νικολάου. Όσο αφορά την εξομάλυνση των σχέσεων με την ε, Κύπρο, και επίσης το πρωτόκολλο της Άγκυρας. Νομίζω ότι ήδη σας έχω καλύψει. Δύο φορές αναφέρθηκα σε αυτό που ρωτήσατε. Και επαναλαμβάνω. Ο θεσμικός μας ρόλος είναι να κάνουμε κάποια αξιολόγηση των πραγμάτων αντικειμενική και μερόληπτη και κατόπιν να αναφέρουμε σχετικά στο Συμβούλιο. Οκτώ κεφάλαια ε, ανεστάλησαν το Δεκέμβριο του 2006 προτάσει δική μας. Πρέπει τώρα να προχωρήσει η Τουρκία να υλοποιήσει το πρωτόκολλο κάτι το οποίο είναι και υποχρεωσή τη και μέτρο οικοδόμηση εμπιστοσύνη. Επίση είχαμε κάποιε ερωτήσει που αναφέρονται στην τουρκοκυπριακή κοινότητα. Το 2004, όπως θα θυμάστε, κατόπιν του δημοψηφίσματος για το σχέδιο ΑΝΑΝ, το Συμβούλιο εκάλεσε την Κομισιόν να υποβάλει προτάσεις ούτως ώστε να βοηθηθεί η επανένωση της νήσου. Και να υπάρξει συνεργασία, ώστε να βοηθεί οικονομικά από την μία πλευρά η άλλη, η τουρκοκυπριακή. 259 εκατομμύρια ευρώ εκταμιεύτηκαν και πρόκειται για μια οικονομική βοήθεια η οποία τρέχει ακόμα και επίσης υπήρξε και συμφωνία ε, απευθείας ελεύθερου εμπορίου μεταξύ της ε, τουρκική κοινότητας και της ε- Ευρώπης πέρασαν πέντε χρόνια ακόμα εκκρεμεί αυτή η απόφαση του ελεύθερου εμπορίου στο Συμβούλιο παρά το ότι το 2007 έγινε και προσπάθεια στο Συμβούλιο όσον αφορά την ε, έγκριση αυτή της πρότασης της Κομισιόν ε, που είχαμε ζητήσει πάλι αμήλυτη να εγκριθεί. Επίσης για να έχετε όλη την εικόνα θα πρέπει και αυτά να τα έχουμε κατά νου. Οπότε ας εστιάσουμε την προσοχή μας στο πώς θα αποσπάσουμε κάποια αποτελέσματα ε, για μια συνολική ρύθμιση του προβλήματος μέσω των διαπραγματεύσεων. Κύριο Κύριλοφ τώρα αναφέρθηκε στο θέμα των θηρήσεων διαβατήριων σε σχέση με την πρώην Ιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας, κύριε Παπα-Νικολάου, πρέπει να σας αναφέρω και σας στο ότι βεβαίω και όλο αυτό το, το μακρινάρι το, το, το αναφέρω και θα ήθελα όμω πάρα πολύ κάποια στιγμή να υπάρχει κάτι πιο εύκολο που να χρησιμοποιούμε. Η χώρα αυτή όμως είναι η κορυφαία, είναι η πρωταθλήτρια όσον αφορά τι επιδόσει των χωρών για να αποσπάσουν την, την άρση των περιορισμών για τα ταξίδια και για τη θεώρηση Άρα θα πρέπει να πιστούμε λοιπόν όλοι ότι υπάρχει ασφάλεια σχετικά με τα ταξίδια εκεί. Όλα αυτά βοηθούν στον να υπάρχει και τη κοινωνία των πολιτών στη χώρα εκείνη. Κύριε Γκέρνε, επίση μα μιλήσατε για την ε, διάβριση σχέση με τη τη Λισαβόνα και αντιλαμβάνομαι από τα επιχειρήματά σα ότι δεν θα αλλάξει τίποτα όσον αφορά τι διατάξει συνθήκε για τη διεύρυνση Άρα θα ισχύουν και όσα ισχύουν σήμερα, ότι δηλαδή οποιαδήποτε ευρωπαϊκή χώρα η οποία σέβεται καποιε αρχέ και τη στηρεί μπορεί να υποβάλει αίτηση ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Επίση, αν κατάλαβα καλά, είπατε ότι μόλι κυρωθεί και τεθεί σε ισχύ η συνθήκη τη Λισαβόνα, τότε μπορούμε να επικεντρώσουμε την προσοχή μα σε κάποια θέματα πολιτική. Πάρα πολύ σωστό είναι αυτό, γιατί τώρα έχουμε διάφορε. Έχουμε συζητήσει σε θεσμικέ σε μια 20 ετία ή τουλάχιστον μια 8 ετία πιο συγκεκριμένα. Οπότε τελικά θα πρέπει να έχουμε κάποια προσωρινά συμπεράσματα όσον αφορά την ε, συνθήκη τη Λισαβόνα Μόλι τη ισχύει, να κάνουμε ό,τι μπορούμε ώστε να ενισχύσουμε την κοινή εξωτερική μα πολιτική. Και να μπορέσουμε ταυτόχρονα να κάνουμε κάτι για την ε, ανάσχεση των συνεπειών της οι μεσονομικές κρίση. Κάποιος άλλο αναφέρθηκε. Α, ναι, στους, για Ρωμάνους. Τι να σας πω γι' αυτό. Το 2004 επί Ολλανδικής Προεδρίας η Ευρωπαϊκή Ένωση έλαβε τη σχετική απόφαση όσον αφορά την προσχώρηση της Βουλγαρίας και Ρουμανίας η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν είχε πιστεί ότι είναι έτοιμη προς η Ρουμανία και θελήσαμε να τάξουμε πλέον προϋποθέσεις ιδίω όσον αφορά δικαιοσύνη και ιστορικές υποθέσεις αλλά και την αναδιάρθρωση του τομέα της Χαλιβουργίας όμως υπήρχε πολιτική πίεση από μεριά των κρατών μελών και οπότε έτσι εμείς ενδώσαμε και αποτέλεσμα ήταν το ότι βάλαμε κάποιες έντρες διαφύλαξεις, ε, η υποπτία ε, αναβαθμίστηκε ε, και οι σχετικές συνέπειες για να πιο αυστηρές όσον αφορά την μη τήρηση των όρων. Και λέγανε οι Ρουμάνοι ότι όλα αυτά είναι καλβινιστική συνωμοσία. Πάρα πολύ. Πάρα πολύ ενδιαφέρον χαρακτηρισμός από θεολογικής πλευράς. Εγώ, ξέρετε, είμαι μέλος της ε, Λουθερανικής Εκκλησίας ε, της Φιλανδίας, αλλά δεν είμαι καλβινιστής. Τέλος πάντων. Και πρέπει και αυτό να το λάβουμε υπόψη. Και στα απομονήματά μου μία μέρα θα σας πω ακριβώς τι έγινε τότε και πόσο βοήθησε η Ολλανδική Προεδρία την ε, προσχώρηση της Ρουμανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα πρέπει να οι θεσμικέ μεταρρυθμίσει σε Βοσνία Ζεγοβίνη. Ε, τώρα αυτά τα θέματα είναι υποδιαπραγμάτευση, δεν μπορώ να σα πω κάτι συγκεκριμένο. Όμω θέλουμε εξέλιξη, όχι επανάσταση όσον αφορά το θεσμικό πλαίσιο για τη χώρα αυτή. Και έχουμε ω αφετηρία την ειρηνευτική συμφωνία του Dayton και θέλουμε το συνταγματικό πλαίσιο της χώρας αυτής να είναι συμβατό με το Ευρωπαϊκό ε, Κοινοτικό Δίκαιο και η χώρα αυτή να συνομιλεί μαζί μας με μία φωνή και επίσης να υπάρχει μία αποδεκτή διαδικασία ε, ένταξη τους, μάλλον μεταφοράς του κοινοτικού δικαίου στο ιστορικό δίκαιο. Αποστολή μας δε αυτή είναι το να εξασφαλίσουμε